Καλημέρα σας. Είναι 9 και 10, νομίζω ότι είναι ώρα να αρχίσουμε και θα αρχίσω να μιλάω τώρα σου παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας. Välkomna Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνεδρίαση. Υπάρχουν αρκετά θέματα επιτάπητο σήμερα. Θα έχουμε και μία σειρά ψηφοφοριών που θα μας πάρουν αρκετό χρόνο. Το πρώτο θέμα βεβαίως είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Και υπάρχει και μία πρόταση αλλαγής στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την γερμηνία, λέει ο πρόεδρος. Όχι, εντάξει, όλα είναι εντάξει. Ωραία λοιπόν, έχει γίνει μια πρόταση τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης. Σήμερα θα, θα είχαμε ψηφοφορία στο σημείο 16 ε, σχετικά με την ε, έκθεση της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ωστόσο, δεν ήταν έτοιμες οι τροπολογίες έγκαιρα, δεν κατέστη δυνατόν να είναι έτοιμες οι τροπολογίες και συνεπώς δεν θα ψηφίσουμε στο σημείο αυτό σήμερα. Αντιθέτως, θα επιτρέψουμε στον εισηγητή να καταθέσει τις δικές του τροπολογίες κατευθείαν. Θα συζητήσουμε λοιπόν την έκθεση της κυρίας Γκόμες, ωστόσο δεν θα ψηφίσουμε. Θα την ακούσουμε να παρουσιάσει τις θέσεις. Μπορούμε λοιπόν να εγκρίνουμε την ημερήθησια διάταξη με αυτήν την τροποποίηση. Ωραία. Ε, 2. Ε, ε, Ωραία λοιπόν, σημείο 2. Πρέπει να σας πω καταρχήν ότι έχουμε μια, ε, ε, την κυρία Μιντούρα Κλεβέτη, η οποία είναι νέα αναπληρωματική, νέο αναπληρωματικό μέλος. Καλώς ήρθατε στην ε, Επιτροπή μας. Η κυρία Κλεβέτη αντικαθιστά την κυρία Πλάμψε. Είναι η πρώτη φορά σήμερα που έρχεται στη συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 4 Ιουνίου, δηλαδή την προσεχή εβδομάδα θα έχουμε μια ανοιχτή ακρόαση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική από τις 3 έως τις 6 το απόγευμα. Τρίτη ανακοίνωση. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν ήδη λάβει μία μελέτη από το Τμήμα Πολιτικής σχετικά με, τις, ε, με τα χαρακτηριστικά του φύλου. Η, στη συνεδρίαση της ΔΕΒΕ στις 18 ε, Ιουνίου από τις 3 έως τις 6 θα λάβετε μία πρόσκληση για συμμετοχή μας εκεί. Επίσης πρέπει να σας πω ότι στις 21 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει μια εκστρατεία, διετή εκστρατεία μάλιστα, με στόχο την συμμετοχή περισσότερων γυναικών στην έρευνα και την καινοτομία για να σπάσουν τα στερεότυπα τα οποία επικρατούν σήμερα όπου δηλαδή οι γυναίκες καταλήγουν να μην έχουν την ίδια συμμετοχή ή τον ίδιο βαθμό συμμετοχής σε αυτόν τον τομέα, την ε, καινοτομία και την έρευνα. Τα μέλη της Επιτροπής θα προσκληθούν να παραστούν στην ε, συνάντηση αυτή στις 21 Ιουνίου. Και ερχόμαστε στο σημείο 3 της ημερησίας διάταξης. Ανακοινώσεις του Προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών. Στους φακέλους σας θα πρέπει να έχετε τα πρακτικά, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις επί των πρακτικών. Προτείνω να εγκρίνουμε τα πρακτικά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, κανένα σχόλιο. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Και ερχόμαστε στο πρώτο ουσιαστικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Och det är kvinnors arbetsvillkor inom Θέμα συνθήκης εργασίας των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών. Η κυρία Περές έχει συντάξει την, ε, την έκθεση και θα δώσω το λόγο αμέσως στην κυρία Περές για να μας παρουσιάσει την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο, αγαπητοί συνάδελφοι. έκθεση που σας παρουσιάζω σήμερα θέτει το θέμα των συνδικών εργασίας των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών είναι ένας τομέας αυτός στον οποίο υπάρχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση του γυναικείου φίλου. Κάνω λοιπόν μια κτηνογραφία των πολλών ζητημάτων που ήδη στο παρελθόν στην Επιτροπή μας εξετάσαμε όπως οι διακρίσεις των τομέα της εργασίας, η διάρκεια των συμβάσεων, συνδυασμός οικογενειακής ζωής και επαγγελματικής, το θέμα της γυάλινης οροφής, όλα αυτά είναι ζητήματα που δυστυχώς βλέπουμε ότι συνεχίζουν να υφίστανται, να επαναλαμβάνονται στην συνήθεια πρακτική σε πολλούς χώρους ε, όπου εξετάσαμε την ε, συνθήκες. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε κάποια σημεία τα οποία κρίνω ότι έχουν την μεγαλύτερη σημασία. Όπως είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι υπάρχει ε, οριζόντιος διαχωρισμός, καταπληρισμός εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη περίπου το ίμιση των γυναικών ασχολούνται με 10 από τα 130 επαγγέλματα της διεθνούς κατανομής ε, επαγγελμάτων. Υπάρχει επίσης μια επικέντρωση της ε, εργασίας των γυναικών στο δημόσιο τομέα όπου εργάζεται το 37% των γυναικών έναντι του 17% των ανδρών. Επίσης ε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η προσωρινή ημερική η μερική απασχόληση είναι μια απασχόληση καθαρά γυναικεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το ζήτημα του ελαστικού αεραρίου είναι κάτι το οποίο γενικεύεται, εργασία τα Σαββατοκύριακα, όλη αυτή, όλη αυτή η ευελιξία και η επιμήκυση του αεραρίου αφορά τις γυναίκες. Ε, τα ωράρια αυτά σημαίνουν ότι δυσκολεύεται η δυνατότητα συνδυασμού της οικογενειακής ζωής και της επαγγελματικής. Επίσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν ε, συγκεκριμένα μέτρα σε αυτόν τον ε, τομέα παροχής υπηρεσιών ε, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην, στα ωράρια με τα οποία ασχολούνται οι γυναίκες γιατί έχουν δυσκολίες στο να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Να πούμε επίσης ότι συνήθως λέγεται ότι οι γυναίκες είμαστε συνηθισμένες να συνδυάζουμε το γεγονό ότι οι άνδρες θα πρέπει να αναλάβουν, να, να συμβιβάζουν συγγνώμη, την ε, οικογενειακή ζωή με την επαγγελματική σε αντίθεση με τους άντρες. Επίσης θέλησαμε να κάνουμε αναφορά στο πλαίσιο της έκθεσης ότι η άνοδος του επίπεδου σπουδών των γυναικών δεν συνέβαλε στην ε, βελτίωση των συνθήκων εργασίας ε, των γυναικών αυτών. Βλέπουμε ότι η συμμετοχή των γυναικών στα πανεπιστήμια είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών. Ε, τα επίπεδα κατάρτισης εκπαίδευση είναι ανώτερα, αλλά δεν συνοδεύονται από μια μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια σε υψηλές θέσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι η γυάλινη οροφή συνεχίζει να υφίσταται και αυτά είναι και αυτά θα πρέπει να διαραγούν ε, έτσι ώστε οι γυναίκες ε, με το κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο να μπορέσουν να ε, δουλέψουν σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Η έκθεση επίσης αναφέρεται στον παραοικονομία και στην κρίση και όσο αφορά τη γενική απασχόληση των μέλων πλησιών, το μέγεθο παραοικονομία είναι μεγαλύτερο από την αντρική απασχόληση, επειδή οι τομεί στου οποίου παραδοσιακά εισέρχονται οι γυναίκε, όπω οι οικιακέ υπηρεσίε, η φροντίδα ατόμων κλπ., χαρακτηρίζονται από μεγάλη απορρίθμιση. αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Η οικονομική κρίση λοιπόν που γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την περίοδο και η απορρίθμιση των ε, συνθηκών εργασίας ε, έχουν ως αποτέλεσμα να καθίσταται όλο και πιο επισφαλή η θέση των εργαζομένων ε, αλλά ιδιαίτερα αυτό συμβαίνει σε κάποιους τομείς όπως οι οικιακές υπηρεσίες. Χρειάζεται λοιπόν ε, να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να νομοθετούν για μια καλύτερη ρύθμιση των ε, οικιακών ε, εργασιών Θέλω επίσης να τονίσω ότι η οικονομική κρίση οδηγεί σε μια επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, στην έκθεση επίσης αναφέρουμε <clears throat> το ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να τροποποιήσει την οδηγία περιμητρότητας, δεχόμενο την ευελιξία που ζήτησε το Ευρωκοινοβούλιο για να προστατευτούν περαιτέρω οι συνθήκες εργασίας ε, των ε, ε, εγγύων γυναικών. Δυστυχώς το ζήτημα αυτό παραμένει εκρεμές εδώ και πολύ καιρό. Το Κοινοβούλιο έκανε ό,τι έπρεπε, προσπάθησε να καταλήξει σε μια θέση κοινή όλων των πολιτικών ομάδων παρετήθηκε από κάποια σημεία τα οποία κρίναμε ότι είναι απαραίτητα, αλλά εμείς τόσο καλός κακός υπάρχει μια θέση του Κοινοβουλίου, χρειάζεται να ζητήσουμε λοιπόν τώρα από το Συμβούλιο να προωθήσει την αποδέσμευση αυτού του φακέλου. Θέλουμε επίσης στην έκθεση να αναφερθούμε στην το θέμα των προσωπικών υπηρεσιών όπως ε, μασάζ ε, κλπ. Θα μπορέσουμε να διευθετήσουμε και το ζήτημα της ε, ε πορνείας αλλά και της εκμετάλλευσης των γυναικών. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν να κλείνουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα Επίσης υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα και καλό τους ε, συναδέλφους ε, να το εξετάσουν. Φυσικά μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η έκθεση με την συνεισφορά των συναδέλφων και σας ζητώ να βοηθήσετε προκειμένου το Κοινοβούλιο να αποφανθεί για επιμίας πραγματικότητας επί τη οποία θεωρώ ότι υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία όχι μόνο στο Κοινοβούλιο μας αλλά και από όλου του δημόσιου θεσμούς. Να καταλήξω ευχαριστώντας ε, για τη συνεργασία του προσωπικού και της γραμματείας. Ε, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Κλέσκα πρώτα απ' όλα. Αναλύοντας ε, την Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας... Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι γυναίκες στον τομέα των υπηρεσιών. Το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό σε αυτόν τον τομέα όσον αφορά τις γυναίκες. Υπάρχουν εδώ τέσσερα βασικά στοιχεία. Η ανισότητα των μισθών, καταρχήν, όπως το γνωρίζουμε, θαυμάσια, η μία από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ίση μισθή για ίση εργασία. Σε ορισμένες χώρες Υπάρχουν τέτοιου ρυθμίσεις, αλλά στην πράξη τα πράγματα είναι διαφορετικά, άλλωστε αυτό το καταδεικνύουν και οι στατιστικέ. Οι γυναίκες έχουν μισθούς χαμηλότερους κατά 16,5% σε σχέση με τους μισθούς των ανδρών. Για παράδειγμα, στην Πολωνία, στον τομέα των υπηρεσιών, οι μισθολογικές διαφορές είναι οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Συνεπώς υπάρχει διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών στην αγορά εργασίας και αυτό το φαινόμενο έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Τώρα, ως προς ε, τον συνδυασμό μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η απουσία υποδομών προκειμένου τα ηλικιωμένα άτομα, τα ηλικιωμένα άτομα και τα παιδιά να έχουν επαρκή φροντίδα και επαρκή προστασία. Οι γυναίκες συχνά αποκλείονται από την αγορά εργασίας για αυτό το γεγονός ακριβώς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ε, και πολύ πιο χαμηλές συντάξεις. Συχνά μία γυναίκα αντί να αναθέσει σε κάποιον άλλον τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των παιδιών, είναι υποχρεωμένη ή μάλλον προτιμάει να εργάζεται λιγότερο για να μπορεί να φροντίζει τα ηλικιωμένα άτομα και τα παιδιά. Η χαμηλή μισθή είναι ένα σημαντικός παράγον εδώ. Βεβαίως, μπορεί να υπάρχουν ε, ελαστικές μορφές εργασίας. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτό ε, είναι θελοντικό. Δεν είναι υποχρεωτικό. Συνεπώς δεν συμφωνώ με την κυρία Περές όσον αφορά ε, το ευέλικτο ωράριο. Η κυρία Περές μας λέει ότι η ευελιξία είναι μειονέκτημα όταν επιβάλλεται δεν είναι κάτι το καλό, αλλά όταν η ίδια η γυναίκα θέλει να έχει ευέλικτα ωράρια, αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο. Τρίτο στοιχείο, οι συνθήκες απασχόλησης. Συχνά οι συμβάσεις εργασίας είναι δεν είναι ευνοϊκέ για τις γυναίκες. Όπως είπε η κυρία Περέζα δικαίως, θα υπάρξουν περισσότερες γυναίκες που θα εργάζονται παράνομα από ότι άντρες. Η κυρία Περέζ έχει δίκιο. Άλλωστε, βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Το τέταρτο στοιχείο είναι ο περιορισμός των θέσεων εργασίας που έχει σχέση με την οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση επηρεάζει πολύ σοβαρά τις γυναίκες και την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και στις υπηρεσίες. Αυτό ε, επηρεάζει και την, την ε, ισότητα δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δυστυχώς, όπως μας δείχνουν τις στατιστικές, η οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες απασχόλησης των γυναικών. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η κατάσταση των ανδρών έχει πολύ επιδεινωθεί. Αλλά οι αναλύσεις καταδεικνύουν ότι οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη ευκολία να επανέλθουν στην αγορά εργασίας από ότι οι γυναίκες. Επίσης, η ιδιομορφία της γυναικείας εργασίας τις βάζει σε δύσκολη θέση επειδή οι γυναίκες εργάζονται κυρίως στο δημόσιο τομέα, ο οποίος υφίσταται αυτή τη στιγμή μεγάλες περικοπές. Η κυρία Περέσε μίλησε για τη θέση της γυναίκας στον τομέα των υπηρεσιών. Ε, μιλάμε για τα στερεότυπα, για τη διακριτική μεταχείριση. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα προκειμένου οι γυναίκες να έχουν μεγαλύτερους μισθούς και να έχουν θέσεις πιο σημαντικές. Πρέπει να υπογραμμίζουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε συχνά συζητήσει. Δηλαδή, ότι η μισθή είναι άνηση για τις γυναίκες και το γεγονός ότι οι γυναίκες κατέχουν πολύ λιγότερες σημαντικές θέσεις από ότι οι άνδρες. Αυτά έχουν σχέση και με το δικαίωμα στη σύνταξη των γυναικών. τα συνταξιδοτικά δικαιώματα συγκεκριμένα. Αυτό αφορά τις γυναίκες που είναι πάνω από 50 ετών. Επίσης, οι γυναίκες δύσκολα προσαρμόζονται στις σημερινές συνθήκες εργασίας, όπου απαιτείται μεγάλη κινητικότητα. Η εργασία των γυναικών στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, της προστασίας των παιδιών, είναι εργασία η οποία δεν αναγνωρίζεται επαρκώς ε, στην κοινωνία. Όταν συγκρίνουμε το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα, στον δημόσιο τομέα υπάρχουν σαφή κριτήρια απασχόλησης. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα η τάση είναι αντίστροφη οι συνθήκες είναι χειρότερες. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ε, στον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Περέζ και θα ήθελα να τη συγχαρώ για την έκθεσή της, η οποία είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και δίνω το λόγο στην κυρία Κόχμεγεν. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τις συζητήσεις μας εδώ, διότι κατορθώσατε να καλύψετε πολλά σημαντικά θέματα που συνδέονται με το θέμα γυναίκες στον τομέα των υπηρεσιών. Νομίζω ότι, όπως επισημαίνετε στην έκθεσή σας, πολλές γυναίκες στην Ευρώπη ε, διακατέχονται από ανησυχία δουλεύοντας στον τομέα των υπηρεσιών, ο στον οποίο κατά κύριο λόγο δουλεύουν οι γυναίκες. Και ασφαλώς ο τομέας αυτός θα αυξηθεί τα προσεχή χρόνια και όλο και περισσότερα άτομα θα ε, εμπίπτουν στο πεδίο ας πούμε ενδιαφέροντος αυτής της έκθεσης. Ενώ συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα αναφέρατε, διότι καλύπτεται πολλά θέματα όπως επεσήμενα, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία τα οποία επιθυμώ να συζητήσουμε, διότι έχω κάπως διαφορετική άποψη. Ε, καταρχήν, ευέλικτες ώρες εργασίας. Νομίζω ότι γενικά Ε, ε, λαμβάνοντας υπόψη την εισαγωγή της έννοιας της ευελιξίας στον χρόνο εργασίας, καταρχήν είναι θετικό αυτό, διότι μπορεί κανείς να συνδυάσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Και είναι κάτι που ε, μπορεί να είναι ελκυστικό και για τους άνδρες οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν αυτό το διπλό ρόλο να συνδυάσουν δηλαδή επαγγελματικές υποχρεώσεις και οικογενειακές. Άρα λοιπόν οι ευέλικτε όλες εργασίες είναι κά... ωράριο εργασίες είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καλωσορίσουμε. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει ένα απλό πλαίσιο, ένα πλαίσιο που θα το καθαστήσει πιο θετικό, πιο ευεργετικό και λιγότερο αρνητικό. Τι σημαίνει, μάλλον η αναζήτηση της ισορροπίας απαιτεί ευελιξία τα παιδιά, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι κλπ. Δεν λειτουργούν ανάλογα με συγκεκριμένα ωράρια. Άρα λοιπόν η ευελιξία γενικότερα ως αρχή είναι μια θετική αρχή. Ωστόσο θα πρέπει να αποφευθεί η κατάχρηση αυτής της δυνατότητας. ευέλικτα ωράρια εργασίας δεν πρέπει να σημαίνει ότι αυξάνει ο όγκος της εργασίας και τούτο νομίζω σημαίνει διάφορες διαχειριστικού περιεχομένου διαδικασίες και θα ήθελα αυτό να το συζητήσω μαζί σας και με άλλους σκιώδες εισηγητές για να αναζητήσουμε μια ισορροπία επ' αυτού. Δεύτερο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω. Όπως ορθώς αναφέρατε, εργασία και οικογενειακή ζωή αφορά κατά κύριο λόγο στις γυναίκες. Είναι αποστολή των γυναικών. Τα πράγματα θα αλλάξουν, πιστεύω, μόνο αν περιλάβουμε στη συζήτησή μας αλλά και στις έκθεσή μας αλλά και γενικότερα στις συζητήσεις μας αν αντιμετωπίζουμε άνδρες και γυναίκες με τον ίδιο τρόπο. Διότι αν συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι είναι θέμα των γυναικών αποκλειστικά θα συνεχιστεί να είναι θέμα των γυναικών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά οι περισσότεροι εξημών θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη αμφότερων των φίλων, ανδρών και γυναικών να εξασφαλίσουν μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και άρα υπάρχει ευθύνη να βοηθήσουμε τους άνδρες, αλλά, ε, τις γυναίκες αλλά και τους άνδρες. Επίσης, όσον αφορά στην ευελιξία και τον αναπτυσσόμενο αυτόν τομέα της οικονομίας, θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις που θα είναι ελκυστικές σε αμφότερα τα φύλλα ώστε να εξασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Διότι τα πράγματα για τις γυναίκες θα αλλάξουν μόνο αν αλλάξουν και τα πράγματα για τους άνδρες. Είμαι πεπισμένη από αυτού. Όσον αφορά στο σημείο 10, αναφέρεται ότι ακόμα λίγες είναι οι γυναίκες οι οποίες συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια. Ε, κάτι το οποίο ε, επικρίνεται πιστεύετε ότι αυτό είναι μια γενικότερη θέση των εταιριών. Και επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι αναφέρατε και πράγματα τα οποία εκ πρώτης όψης δεν είναι και τόσο προφανή. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την έκθεσή σας. Η κυρία Κλεβέτη έχει τώρα το λόγο. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Περέζ αυτό είναι ένα μόνιμο πάγιο θέμα θα έλεγα στις συζητήσεις των επιτροπών όπως τη δική μας. Αλλά ποτέ δεν έχουμε πει αρκετά διότι δεν πρέπει να λησμονούμε ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα που δεν έχουν βρει ακόμα τη λύση τους. Αυτό το οποίο μας πρότεινε προς συζήτηση η κυρία Περέζη είναι κάτι το περίπλοκο. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να επιμείνω πάνω στο θέμα ε, του συνδυασμού της οικογενειακής ζωής ε, με την επαγγελματική ζωή. Το σημείο 15 μας λέει ότι καταρχήν πρέπει να ενθαρρύνουμε, να λάβουμε μέτρα ώστε αυτό να πραγματοποιηθεί στον κόσμο. Αλλά αυτό αφορά και τις γυναίκες και τους άντρες. Το γεγονός όμως παραμένει ότι οι γυναίκες είναι εκείνες ε, οι οποίες θεωρούν αφενός ότι είναι καθήκον τους να βοηθήσουν περισσότερο την οικογένεια, να φροντίσουν τα παιδιά και τα λοιπά. Γιατί στη χώρα μου, στη Ρουμανία, εάν μιλήσει κανείς με τις γυναίκες, θεωρούν ότι αυτό είναι ο καθήκον τους. Αυτό όμως δεν είναι σωστό, διότι πρέπει να επιμείνουμε οι άντρες και οι γυναίκες σε μια οικογένεια ε, να μοιράζονται τις ευθύνες, να υπάρχει ισότητα όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών, για παράδειγμα αλλά το γεγονός παραμένει ότι η γυναίκα είναι εκείνη η οποία αναλαμβάνει περισσότερο από τον άντρα αυτή την ευθύνη του συνδυασμού, δηλαδή ε, της επαγγελματικής με ε, την ε, προσωπική ζωή, με την οικογενειακή ζωή. Και τα τελευταία χρόνια οι νέες γυναίκες που έχουν παιδιά δείχνουν ότι τα καταφέρνουν, προσπαθούν να τα καταφέρουν. Γι' αυτό πρέπει να τις ενθαρρύνουμε και πρέπει να τις βοηθήσουμε με συγκεκριμένα μέτρα για να τα καταφέρουν. Παράλληλα όμως πρέπει και οι άνδρες, όπως είπε η συνάδελφος, και εκείνοι, και οι άνδρες δηλαδή, να αντιληφθούν ότι τα ίδια καθήκοντα πρέπει να τα μοιράζονται και εκείνοι. Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονούμε τις μονογονεϊκές οικογένειες που κατά κανόνα ε, απαρτίζονται από τη γυναίκα και τα παιδιά και δεδομένου το διαζύγιο είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πολύ εύκολα σήμερα. Και επειδή υπάρχουν οικογένειες όπου δεν υπάρχουν ε, ζευγάρια υπό την επίσημη μορφή, υπάρχει, αν θέλετε, κινητικότητα και στον τρόπο που διαμορφώνεται η οικογένεια, πάλι τελικά η γυναίκα είναι εκείνη που αναλαμβάνει τις μεγαλύτερες ευθύνες. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι το σημείο 15 να το υπογραμμίσουμε, να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Επειδή δεν πρέπει απλώς να πούμε ότι το ιδανικό είναι να συνδυάζεται η οικογενειακή ζωή με την επαγγελματική ζωή. Δεν πρέπει να είναι μόνο ένα ιδανικό. Πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες επειδή μπορούμε να μελετάμε το θέμα, να τοποθετηθούμε πάνω στο θέμα, αλλά οι οικογένειες είναι εκείνες που πρέπει να βρουν ε, το πιο δίκαιο τρόπο ε, μεταξύ των συντρόφων συζύγων ε, για να φροντίσουν τα παιδιά τους. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να προτείνουμε συγκεκριμένα μέσα διότι το 2050 πάλι θα συζητάμε για την, τον συνδυασμό, τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού ε, βίου. Σταματάω εδώ ε, λέγοντας ότι υπήρξα μέλος της Κοινοβουλικής Συνέλευσης της Συμβουλής Ευρώπης επί 8 χρόνια και το πρόβλημα του συνδυασμού της οικογενειακής ζωής με την επαγγελματική ζωή είναι ένα θέμα που απασχολεί και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, θα μπορούσαμε λοιπόν να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο της Ευρώπης για να βρούμε ίσως νέες ιδέες. Εδώ όμως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε συγκεκριμένες και σημαντικές λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Γέροκα να έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Είναι εξαιρετικά καλή η έκθεσή σας κυρία Πέρες επειδή είναι σύνθετη και δείχνει ακριβώς την ε, ευρεία συνεισφορά των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ε, όλα αυτά τα εμπόδια, τα προσκόμματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονιστεί η παρούσα κατάσταση κρίσης που καθιστά τις γυναίκες, μάλλον που φέρνει τις γυναίκες σε ακόμα πιο τρωτή και ευάλωτη θέση, που ούτως ή άλλως είναι θύματα ανισότητας στον τομέα των υπηρεσιών. Πρόσφατα το Συμβούλιο ενέκρινε ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ουσιαστικά είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Γυναίκες και αφορά περίπου 20 εκατομμύρια γυναίκες. 40% εξ αυτών δουλεύουν στη μαύρη αγορά, στη μαύρη αγορά εργασίας. Και το σύστημα δεν τις αναγνωρίζει, δεν τις, μάλλον δεν τις, δεν τις γνωρίζει, δεν την ξέρει. Και ε, ε, ισχύει αυτό ε, και στις 27 χώρες. Δεν ξέρουμε σε τι βαθμό οι χώρες το γνωρίζουν. Τα προγράμματα είναι πολύ περιορισμένα και όλες οι συστάσεις που κάνετε στην έκθεσή σας είναι εύστοχες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτές τις γυναίκες, γιατί όπως λέτε και στην έκθεσή σας, αυτές είναι γυναίκες από, που ανήκουν σε μειονότητες ή γυναίκες από μόνο γονεϊκές οικογένειες και όλες αυτές είναι εξαιρετικά ευάλωτες. Από την άλλη υπάρχουν τεράστιες ε, εθνοτικές, εθνικές διακρίσεις σε αυτόν τον τομέα των υπηρεσιών. Τα σημεία που ε, εστιάζετε στην έκθεσή σας και τα στοιχεία που μας δίδετε πραγματικά επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι πάνω από 20 εκατομμύρια Ευρωπαίες γυναίκες βρίσκονται σε αυτή την εξαιρετικά δυσάρεστη θέση. Θα ήθελα λοιπόν να σας συγχαρώ για το περιεχόμενο, το σύνθετο περιεχόμενο της έκθεσής σας. Ο Πρόεδρος ευχαριστώ. Η κυρία Τσούμπα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να πω ότι αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική έκθεση. Ένας ε, πολύ μεγάλος αριθμός ε, ανθρώπων, γυναικών συγκεκριμένα δουλεύουν στον τομέα των υπηρεσιών και άρα είναι εύστοχο να συνταχθεί μία έκθεση για την ιδιόμορφη θέση που βρίσκονται οι γυναίκες αυτές. Πρέπει να πω ότι ως ομάδα θα καταθέσουμε σειρά τροπολογιών. Θα ήθελα να περιγράψω απλώς τη θέση μας όσον αφορά στην ευελιξία. Ε, το ευέλικτο ωράριο εργασίας δηλαδή. Αυτό είναι ένα κυρίαρχο θέμα το οποίο προκύπτει όταν συζητούμε τον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς βλέπουμε τα πράγματα είναι το εξής. Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα αγορά εργασίας, η ευελιξία δεν εφαρμόζεται προς το συμφέρον των γυναικών ή των εργαζομένων ε, γενικά. Συνήθως αυτή η των εργαζομενων γενικα συνηθως αυτη η ευκαμψία εξυπηρετεί τους εργοδότες. Αυτή είναι η κατάσταση στην αγορά που σήμερα γνωρίζουμε. Δηλαδή, το ευέλικτο ωράριο εργασίας δεν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις επιλογές και την επιθυμία των ε, γυναικών, αλλά εφαρμόζεται σύμφωνα με τις επιταγές των εργοδοτών. Συνεπώς, ε, ασφαλώς πρέπει να προστατέψουμε τις γυναίκες. Θα πρέπει να είναι δυνατό οι γυναίκες να ζητούν ευελιξία, για να μπορούν να συνδυάσουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Αλλά τι βλέπουμε μπροστά μας στον πραγματικό κόσμο. Βλέπουμε αυτούς που μιλούν υπέρ της ευελιξίας ε, ουσιαστικά θέλουν να ε, απαλείψουν στοιχειώδεις εγγύησης εργασίας που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι υπέρ και προς το συμφέρον των εργαζομένων αυτές οι απαιτήσει. Άρα λοιπόν γενικώ συμφωνούμε με αυτά που περιλαμβάνεται στην έκθεσή σας, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να εισαχθούν και κάποια άλλα πράγματα για να καλυφθεί ακριβώς αυτός ο σύνθετος χαρακτήρας του θέματος. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Εγώ τώρα θα, θα λάβω εγώ το λόγο στη σειρά των ε, ομιλητών. Το θέμα το οποίο ετέθη νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Οι συνθήκες Όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας, τουλάχιστον στη δική μου χώρα, υπάρχει ένα θέμα με τη μερική απασχόληση. Οι γυναίκες προτιμούν τη μερική απασχόληση και αυτό και στην τοπική αυτοδιοίκηση Ε, ε, ωστόσο γίνονται και πολύ περίεργες ρυθμίσεις και διαπιστώνει κανείς ότι μια γυναίκα η οποία κάνει την επιλογή της μερικής απασχόλησης ουσιαστικά δεν δουλεύει 97% φορές και δουλεύει 3%. Άρα λοιπόν η διευθέτηση αυτή πρέπει να γίνει με πιο ορθολογικό τρόπο. Δηλαδή δεν πρέπει να εξαναγκάζονται οι άνθρωποι, οι γυναίκες συγκεκριμένα, να δουλεύουν υποκαθεστώς μερικής απασχόλησης. Διότι με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η οικονομική ανεξαρτησία αλλά και οι προοπτικές μελλοντική καλύτερης εργασίας. Σκεφτήκατε τι μπορούμε να κάνουμε πιο συγκεκριμένα στις χώρες μέλη για να ε, ε, λύσουμε ή να υπερπηδήσουμε αυτό το πρόβλημα. Αν εξετάσουμε τους τομείς όπου δουλεύουν ε, κατά κύριο λόγο άνδρες, αυτό το πρόβλημα δεν υφίσταται. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα υφίσταται σε δουλειές όπου κατά κύριο λόγο απασχολούνται γυναίκες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να εξετάσουμε. Κύριε Παπαδοπούλου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω έγινε μια αγώνιμη συζήτηση. Θα συγχαρώ και εγώ τη συγγραφέα για την έκθεσή της, γιατί είναι περιεκτική και περιλαμβάνει όλα όσα θα έπρεπε να συμπεριληφθούν. Να επισημάνω ότι ε, στη δική μου χώρα οι γυναίκες κυρίως θέλουν να εργοδοτηθούν στο δημόσιο τομέα, αλλά και στον τραπεζικό τομέα, γιατί ακριβώς τα ωράρια εργασίας είναι καλύτερα ε, στο δημόσιο τομέα εργάζονται μέχρι τις 2.30 ώρα, ενώ στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να εργάζονται μέχρι τις 6 το απόγευμα. Επομένως, είναι ένα κίνητρο να επιδιώκουν εργασίες που να τους παρέχουν την ευχαίρεια να έχουν ελεύθερο χρόνο και να συνδυάζουν επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Και εδώ ακριβώς είναι που πρέπει το ίδιο το κράτος Στι 27 χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έρχεται άρωγος. Γιατί εμεί ω γυναίκε μέλη τη Επιτροπή επισημαίνουμε τα ίδια πράγματα σε όλε τι εκθέσει. Όμω θεωρώ ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει μια ε, διαδικασία ώστε να εναρμονίσει τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το κράτο παρεμβαίνει και βοηθά έμπραχτα στη συμφιλίωση των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Και διευκρινίζω χρειάζονται να υπάρχουν υποδομές φροντίδας των ηλικιωμένων ατόμων, των παιδιών, των βρεφών. Εάν αυτό αναλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα, συνήθω συνεπάγεται πολύ ψηλέ ε, τιμέ που δεν είναι προσιτές για τα βαλάντια των σημερινών γονιών και των οικογενειών λόγω και τη οικονομική κρίση. Επομένω, η δική μου εισήγηση για να είμαστε πρακτικοί είναι ότι σε τέτοιε εκθέσει θα πρέπει να επισημαίνεται η σημασία του gender budgeting όταν καθορίζονται οι εθνικοί προπολογισμοί τι κονδύλι θα δίνεται από το ίδιο το κράτος αλλά και από ευρωπαϊκά προγράμματα στο να ενισχύονται ακριβώς οι υποδομές φροντίδας για τους ηλικιωμένους, για τους μονογονιούς και για τη φροντίδα των βρεφών και των παιδιών. Κάτι τέτοιο έμπρακτα θα στηρίξει τη συμφιλίωση οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων και νομίζω πρέπει να υπάρχει μια αναφορά στο gender budgeting. Και το δεύτερο σημείο, το οποίο θα ήθελα να ενισχυθεί στην έκθεση, είναι ακριβώς αυτό το ψηφιακό χάσμα το οποίο υπάρχει. Οι γυναίκες, αν εξαιρέσουμε αυτές που είναι καλά μορφωμένες και έχουν δύο και τρία πτυχία, σίγουρα γνωρίζουν να χρησιμοποιούν και το διαδίκτυο και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όμως σε πολλές χώρες τις πλατιές μάζες των γυναικών το διαδίκτυο ε, είναι κάτι απόμακρο και ο ηλεκτρονικός αλφαβητισμός, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός υπάρχει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ειδικά προγράμματα εκμάθησης ακριβώς της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή γιατί αυτό είναι ένας πρακτικός τρόπος για να μπουν περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας και να ζητούν ψηλά πόστα και καλύτερες συνθήκες εργοδότησης. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ. λέει ο Λοιπόν, θέλει η κυρία Πέρας να απαντήσει ή να δώσω πρώτα το λόγο στην Κομισιόν καλύτερα ε, και να απαντήσετε μετά. Τι θέλετε, να ακούσετε την Επιτροπή θέλετε. Ωραία. Ωραία τότε παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν εκπρόσωπός της είναι εδώ, να λάβει το λόγο, να μας πει δύο λόγια. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν ε, συμφωνεί με την ε, έκθεση που αφορά στον ε, εργασία των γυναικών για την επισφαλή εργασία, χαμηλή αμοιβή κλπ. Η Κομισιόν τονίζει τις ανισότητες που υπάρχουν ε, ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες σε αυτόν τον τομέα, κάτι το οποίο δημοσίευσε πρόσφατα. μια, σε ό,τι φορά μια πρωτοβουλία για την ε, αύξηση της ε, απασχόλησης, η Κομισιόν ανέλαβε μια αντιμετώπιση τομεακή. Ε, Επίση ε, έχει προτείνει ένα πρόγραμμα για την πράσινη οικονομία για του εργαζόμενου στον τομέα τη ε, υγεία μια ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα των ΤΙΚ. Η Κομισιόν προτείνει να υπάρξει διαβούλευση σε ό,τι αφορά την απασχόληση ποιότητας. Αυτή η ανακοίνωση υπογραμμίζει τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και των ε, χαμηλές αμοιβές στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών. Και το σύνολο των κλάδων η ανακοίνωση της Κομισιόν προτείνει να εγγυηθούμε αμοιβέ ε, ε, βιώσιμε την καταπολέμηση της ανεργίας και να εγγυηθούμε τις Συνθήκε για την καταπολέμηση του κατακαιρματισμού της αγοράς εργασίας. Ε, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα Ανδρογυναικών προτείνει μια σειρά δράσεων συγκεκριμένων όπως τόνισε και η συγγήτρια στην έκθεσή της. Π.χ. η εκπροσώπηση των γυναικών στον τομεί ε, λήψη απόφαση, στον συνδυασμό τη προσωπική, ε, οικογενειακής και εργασιακή ζωής ε, και επίσης εμείς θέλουμε να συμπεριλάβουμε την στρατηγική του φίλου στην, ε, την ε, διάσταση του φίλου στη στρατηγική 2020 Κομισιόν τονίζει την αύξηση της συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασία που θα συνοδεύεται και από τα κατάλληλα φορολογικά μέτρα δομές, υποδομές υποδοχής των παιδιών και την καταπολέμηση σε την διαφορετική αμοιβή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Πέρες για να απαντήσει. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την συμβολή στη συζήτηση. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και τέθη επιτάπητος όχι μόνο το ζήτημα του προβληματισμού επί των επιμέρους ζητημάτων που θέσαμε, αλλά να δούμε και την πραγματικέ δυνατότητε που υπάρχουν για το Ευρωκοινοβούλιο και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ο πρόεδρο είπε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια νομοθετήματα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια ζήτηση πολύ ευρύτερη από ότι αυτή που αφορά τι γυναίκε στον τομέα των υπηρεσιών. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αυξήσουμε την εναρμόνιση των νομοθεσιών των εθνικών σε ζητήματα εργασιακά. Κατά την άποψή μου, ναι, δεν ξέρω αν η στιγμή είναι καταλληλότερη για να υπάρξει παρόμοια πρόοδο, αλλά όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία που έχουν τεθεί με τη συζήτηση. Τώρα, σε ό,τι φορά την ευελιξία, Κατανοώ ότι το θέμα αυτό θα προκαλέσει συζητήσει, αλλά έχει σημασία να συνεχίσουμε να το τονίζουμε. Ίσως να πρέπει να βρούμε μια καλύτερη διατύπωση της παραγράφου που θίγει το ζήτημα της ευελιξίας, αλλά συμφωνώ 100% με την συνάδελφο Σούμπερ, Δηλαδή η ευελιξία ε, όταν είναι ε, απαραίτητη για να προσαρμοστούν στις ανάγκες ε, των εργαζομένων είναι κάτι το θετικό φυσικά. Αλλά το ζήτημα είναι πως οι εργασιακές νομοθεσίες θέτουν αυτή την δυνατότητα προς το μέρος αυτού που διαπραγματεύεται τις συνθήκες. Να θέσω ένα παράδειγμα για να γίνω καλύτερα κατανοητή. Ε, έχουμε έναν άντρα εργαζόμενο που θέλει να συνδυάσει την ε, προσωπική ζωή με την εργασιακή. Θέλει λοιπόν να έχει μια δουλειά 20 ώρες περίπου την εβδομάδα και έτσι να μπορέσει να συνδυάσει το ζήτημα της ανατροφής των παιδιών του. Εντάξει, 20 ώρες εβδομαδίως. Τις Δευτέρες όμως ε, θα δούμε, λέει ο εργοδότης, πώς θα γίνει αυτή η κατανομή των ερών. Τη μία μέρα θα έρθει 7 ώρες, ε, άλλη μέρα θα έρθει 2, την επόμενη 7. Την επόμενη εβδομάδα όμως αλλάζει άρδιν αυτή η κατανομή. Μα αυτή είναι ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί αδυναμία στον εργαζόμενο να συνδυάσει την εργατική, την, την εργατική ζωή με την ε, οικογενειακή. Και έτσι βλέπουμε λοιπόν πώς μπορεί να επηρεάσει ο περίφημος όρος ευελιξία στην την πραγματικότητα των εργαζομένων. Πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη διατύπωση λοιπόν πέρα αυτό είναι σίγουρο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ελπίζω πως με τις ε, συμβολές των συναδέλφων θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω το κείμενο. Είμαι στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε και να βελτιώσουμε κατακλείδη το κείμενο μετά από τα όσα ακούσαμε στο πλαίσιο της συζήτησης που είχαμε σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και ευχαριστώ τους πάντες για τη συζήτηση. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 6η Ιουνίου το μεσημέρι. Η Επιτροπή θα ψηφίσει τα... στις 10 Ιουνίου και αυτή θα είναι η τελευταία μας συνεδρίαση πριν από τις θερινές διακοπές και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο. Ε, κλείνει. Τελειώνουμε λοιπόν με το σημείο αυτό και υπάρχει μια ελαφρά αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Συνεπώς θα ασχοληθούμε με το σημείο 6 πριν από το σημείο 5. Εντάξει. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε το χρόνο σωστά ώστε να ασχοληθούμε και με το σημείο 5 αμέσως μετά. Κοινέ διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και κατάργηση του κανονισμού. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ζούμπερ, η οποία είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. De, de parecer que, que apresentamos em relação ao novo regulamento. Η γνωμοδότηση που έχετε αναχείρα σχετικά με τον νέο κανονισμό για τα ταμεία είναι μια πρόταση η οποία στοχεύει στο να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών και αυτό στο πλαίσιο της ε, σημερινής ε, κρίσιμης συγκυρίας κρίση η οποία πλήττει τις ε, γυναίκες πολύ πιο έντονα Θεωρούμε λοιπόν πως ε, σε περίοδους οικονομικής κρίσης, ε, σε περίοδους ε, υποχώρησης των κοινωνικών, εργασιακών και οικονομικών δικαιωμάτων, έχει ιδιαίτερη σημασία να μην περιοριστούν οι χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις ή στην περίοδο κρίσιμη είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι επιδοτήσεις θα πρέπει να αυξηθούν ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους, πιο ευάλωτους τομείς. Γνωρίζουμε ότι για βασικές ανάγκες ε, και ζητήματα όπως το θέμα της απασχόλησης ε, διακυβεύονται θέσεις εργασίας και τότε όλα τα δικαιώματα τα οποία άπτονται της ισότητας διακινδυνεύουν διότι μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Εμείς δεν θέλουμε όμως να ξεχαστούν αυτοί οι πυλώνες, αυτά τα λάβαρα τα οποία μας οδήγησαν στην πρόοδό μας και την οικονομική εφημερία στην οποία έχουμε επιτύχει. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό δεν πρέπει να υποχωρήσουμε επειδή αντιμετωπίζουμε οικονομικές δυσκολίες. Λοιπόν, εμείς αυτήν την γνωμοδότηση που έχετε αναχείρες αναφερόμεθα σε κάποια σημεία. Πρώτα απ' όλα ε, τονίζουμε ότι οι προτεραιότητες ε, των ταμείων θα πρέπει να τονίζουν την ε, αρχή της ισότητας μεταξύ άνδρων και γυναικών. Επίσης ε, τονίζουμε την ε, ισότητα των φύλων και να έχουμε στοιχεία αναλυτικά αναφύλων στις ε, διάφορες φάσεις χρηματοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα στοιχεία να ε, υποβάλλονται αναλυτικά, ειδικά όταν μιλάμε για εταιρική σχέση και για θέματα που άπτονται των στρατηγικών οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν. Επίσης τονίζουμε και την ε, εποπτεία, την επιτήρηση αυτών των προγραμμάτων. Αναφερόμαστε σε κάποια θέματα Ειδικά με την εταιρική σχέση και την συμπερίληψη σε αυτές ε, τις οργανώσεις για την προστασία των δικαιωμάτων γυναικών. Ε, και κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να τονίσω, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. πρέπει να την υπόψη το γεγονό ότι η επιστήμη βοήθεια θα περάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ως αυτού θα θέλαμε το ταμείο αυτό να λάβει περαιτέρω χρηματοδότηση. Επειδή θα αναλάβει αυτή την επιπλέον αρμοδιότητα, αυτή τη νέα αρμοδιότητα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, θα πρέπει να προβλεφθεί ε, μια αύξηση της πρικοδότησης ε, του Κοινωνικού Ταμείου. Διαφορετικά δεν ε, θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις, στους ε, στόχους του. Και άρα θα μπορέσει να παρέχει την ε, απαραίτητη εμπιστητική βοήθεια. Και ειδικά σε αυτή την περίοδο όπου θα έπρεπε να ενισχύσουμε τις δυνατότητες αυτές επειδή υπάρχει αύξηση της ένδυας στην Ευρώπη, αύξηση της φτώχειας των εργαζομένων γενικότερα. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η δράση, αυτή η αύξηση της πρικοδότησης είναι απαραίτητη. Και κάτι ακόμα το οποίο δεν άπτεται αποκλειστικά των γυναικών, να αναφερθώ σε ένα άλλο στοιχείο. Σε όλες τις υπηρεσίες ε, επιστημικής ε, βοήθειας, ε, γενικότερα βοήθειας ε, προς ε, πρόσωπα τα οποία αντιμετωπίζουν δύσκολες ε, συνθήκες. Υπάρχουν οι γυναίκες συχνά είναι αυτές οι πιο θαραλέες που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που γνωρίζει ο πληθυσμός μας. Είναι και αυτό το στοιχείο που εμπίπτει στο πλαίσιο της προβληματικής. Δεν μιλάμε λοιπόν για βοήθεια σε τρόφιμα, μιλάμε για, ιδιαίτερα για γυναίκες και κάτι ακόμα προτείνουμε την διαχωρισμό της αρχής της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό ως πολιτική ομάδα. Διότι πιστεύουμε στην δυνατότητα διακοπής ε, των πόρων για, σε κάποιες χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Τώρα η διακοπή, η ανάκληση αυτής της βοήθειας ε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να συμβεί, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο. Η αλληλεγγύη είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε συχνά. Ακριβώ λοιπόν στην περίοδο αυτή που κάποιες ε, κράτη αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα έντονα, αυτή η βοήθεια θα πρέπει να αυξηθεί, να ενισχυθεί για να προαχθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση και η ισότητα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κράτσα έχει το λόγο. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την ε, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής μας διότι ανέδειξε ε, το ρόλο που μπορεί να παίξουν τα διαφορετικά ταμεία στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά στην ε, ε, δημιουργία συνθήκων για να μπορέσουν οι γυναίκες να αντιμετωπίσουν τις διακρίσεις και να παίξουν τον ρόλο τους στην κοινωνία και στην οικονομία. Ε, συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να είναι σαφές στις αρχές των ταμείων η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ε, και οι πόροι να κατευθύνονται ε, σε δράσεις που ακόμη έχουμε ανάγκη για την ε, ισότητα των γυναικών. Επαναλαμβάνω, από τη μια μεριά για να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις και από την άλλη για να δώσουμε νέες ευκαιρίες στις γυναίκες. Ε, συμφωνώ επίσης ότι το θεωρώ πολύ επιφανειακή, τιμωρητική και όχι αναπτυξιακή και δίκαιη την πρόβλεψη να σταματάτε η χρηματοδότηση σε χώρες με, με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έχουμε πολλά εργαλεία έχουμε υιοθετήσει πρόσθετα εργαλεία μέσα στο πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχία, μέσα από άλλους μηχανισμούς, ούτω ώστε να συμμορφώνονται έγκαιρα οι χώρες και να μην ε, ε, θεωρούμε ότι με την ε, διακοπή της χρηματοδότησης ε, κάνουμε το καθήκον μας. Αντίθετα θα πρέπει να προβλέψουμε το ώστε η χρηματοδότηση να πηγαίνει σε σωστές κατευθύνσεις, να γίνεται σωστή αξιολόγηση της απορρόφησης, του impact της απορρόφησης στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία και όχι την εύκολη λύση της διακοπής. Ε, αν και αυτό δεν άπτεται ιδιαίτερα της ε, Επιτροπής μας. Είναι μια ευρύτερη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η συγγήτρια, ότι και θα είναι και το πνεύμα των τροπολογιών που θα καταθέσω, ότι ε, πρέπει να φροντίσουμε οι γυναίκες να είναι μέσα στις διαδικασίες. Ε, παραδείγματος χάρη εκεί που προβλέπεται μια, η, συμμετοχή εκεί που προβλέπεται η Εθνική Επιτροπή που συνεπικουρεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι αρκεί να υπάρχει μόνο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρέπει και εκπρόσωπος του φορέα α, ισότητας της κάθε χώρας. Πρέπει να υπάρχει ένα μάτι δηλαδή εκεί ε, ε, που ε, επιμελείται την ένταξη και την εφαρμογή της γυναικείας διάστασης. επίσης πρέπει να σημειώσουμε σημειώσουμε ιδιαίτερα ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε και την γυναική επιχειρηματικότητα. Αν μιλάμε για ανάπτυξη, για θέσεις εργασίας, μιλάμε για δημιουργία επιχειρήσεων. Άρα, επειδή έχουμε ψηφίσει πολλές φορές και γνωμοδοτήσεις και τροπολογίες και εκθέσεις όπου ε, τονίζουμε τη σημασία της γυναικείας επιχειρηματικότητας, νομίζω ότι το ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει και να εκπαιδεύσει γυναίκες για αυτές, για αυτή την επιχειρηματικότητα και να βοηθήσει τις γυναίκες να, να κάνουν βιώσιμες επιχειρήσεις. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ε, παρατηρείται γενικά ότι οι γυναίκες έχουν έλλειψη επι, ε, ενημέρωσης και πρόσβαση στην ενημέρωση. Και οι ίδιες το ψάχνουν λιγότερο να ενημερωθούν για τα τρέχοντα, για τις ευκολίες αξιοποίησης των διαθροτικών ταμείων, αλλά και οι φορείς, οι επιχειρηματικοί, οι συνδικαλιστικοί ε, λιγότερο έχουν την έννοια να ενημερώσουν τις γυναίκες. Λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να φροντίσουμε και αυτό, τους διάβλους ε, πληροφόρηση των γυναικών για τα δικαιώματά τους και για τις ευκαιρίες που εμπεριέχονται στα διαφορετικά ταμεία και επίσης στους δείκτες αποτελεσμάτων ε, νομίζω ότι πάσχουμε στην αξιολόγηση ε, και, στις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και την κοινωνία. Στους δείκτες λοιπόν αξιολόγησης πρέπει επιμελώς να λαμβάνεται υπόψη η γυναικεία διάσταση. Αυτές είναι έτσι οι γενικές μου παρατηρήσεις και συμβολή στη γνωμοδότησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ την κυρία Μάιλες από την Επιτροπή αν θέλει να μιλήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια σχετικά με δύο ή τρία σημεία που θίξατε και στο σχέδιο χρονομοδότησης. Καταρχήν θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η Επιτροπή πιστεύει ότι η ισότητα των φύλων είναι μια σημαντική οριζόντια αρχή. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε στα, στις αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού των κοινών διατάξεων υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο υπογραμμίζει ότι οι εταιρικέ σχέσει πρέπει να περιλαμβάνουν φορεί που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση τη ισότητα και τη μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των μερών στι ε, στις συμβάσεις και υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι σε όλα τα στάδια της υλοποίηση ο στόχος πρέπει να είναι να, να εξαλειφθούν οι ανισότητες και θα πρέπει να προωθηθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στι αιτιολογικέ σκέψει αναφέρονται αυτά. Και σε ένα από τα άρθρα επίση υπογραμμίζουμε το γεγονό ότι τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση των θεμάτων ισότητας προωθείται στην προετοιμασία καθώς και στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι περιττό να προσθέσουμε οτιδήποτε άλλο, δεδομένου ότι για μας είναι μια σημαντική οριζόντια προτεραιότητα. Νομίζω ότι αυτό αρκεί. Επίσης, υπάρχει ε, η, η, εξάντε, η προϋποθέση εξάντε για την ισότητα ε, των φύλων και τη διακριτική μεταχείριση. Αλλά λυπούμεθα που το Συμβούλιο δεν συμφώνησε. Και αυτό όμως θα θέλαμε να το θέσουμε υπόψη σας, είναι κάτι το οποίο περιλάβαμε στον κανονισμό. Ως προς τους δείκτες γενικά, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τους δείκτες, αλλά όσον αφορά την κατανομή αναφύλω για ε, τους δείκτες, σύμφωνα με την πείρα μας, πιστεύουμε ότι αυτό δεν αρκεί πάντοτε. Συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση όταν είναι κάτι το λογικό για όλους τους σχετικούς δείκτες. Αλλά πιστεύουμε ότι είναι επίσης σημαντικό να γίνονται αξιολογήσεις και μελέτες για να δούμε ποια είναι η κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη. Και επίσης τα διάφορα κράτη-μέλη ξεκινάνε από διαφορετική θέση. Γι' αυτό δεν θα θέλαμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα υπάρχει μια γενική προσέγγιση, ένα πρόγραμμα, ένα πρώτο πρόγραμμα με κατανομή, με δείκτες που θα κατανέμονται αναφύλλο. Πρέπει να τα δούμε με μεγαλύτερη προσοχή. Νομίζω ότι οι δείκτες δεν αρκούν, θα πρέπει να συνοδεύονται και από κάτι άλλο. Και όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε, τόσο το καλύτερο φυσικά. Ως προς την οικονομική διακυβέρνηση και ε, και οι μακροοικονομικέ τα ταμεία του κοινού στρατηγικού πλαισίου μπορούν να επιτύχουν μόνον εάν υπάρχουν υγιείς δημοσιονομικέ πολιτικές που οδηγούν στην ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι οι εθνικέ κυβερνήσεις θα πρέπει να χαράξουν τις ορθές πολιτικές και να προβούν στις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να υπάρχει η καλύτερη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων των ταμείων. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε τη διασύνδεση μεταξύ ε, των ταμείων του ΚΠΣ και του νέου μηχανισμού της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Κλέβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πιστεύω κράδαντα στις πολιτικές ισότητας, διότι ε, εξασφαλίζει το ελάχιστο επίπεδο κάθε μορφής διακυβέρνησης και αυτό το επίπεδο είναι οι περιφέρειες και σε μια εποχή πολύ περιορισμένων δημοσιονομικών όπου όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν την χρηματοοικονομική κρίση, αυτός είναι ένας τρόπος να βοηθήσουμε όχι μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, την έρευνα, ε, τον τομέα των μεταφορών και όλους εκείνους τους ε, τομείς οι οποίοι εμπεριέχουν το στοιχείο της ισότητας ευκαιριών των δύο φύλων. Έτσι λοιπόν, συζητώντας το κοινό στρατηγικό πλαίσιο ένα από τα πρόσφατα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η έλλειψη η μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Αυτό θα πρέπει να καταγραφεί υπό τη μορφή που έχει και δουλεύουμε εναντίον αυτού, διότι δεν υπάρχουν αναλύσεις που μας δείχνουν ότι θα υπάρξει κάποια διαφορά ε, αν εφαρμοστεί αυτή η μορφή μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Αν θέλει κανείς να δρομολογήσει νέες πολιτικές θα πρέπει να το κάνει στο απόλυτο επίπεδο βάσης, στο τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγήτρια που το περιέλαβε αυτό στην έκθεση. Νομίζω ότι η έκθεση ως έχει αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά καλή. Πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά ζητήματα έχουν περιληφθεί και ιδιαίτερως η αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ένα από τα ε, ταμεία που στο επόμενο πλαίσιο 2015-2020 θα είναι αυτό το οποίο θα ε, πληγεί περισσότερο ενώ από την άλλη οι ανάγκες, ε, οι ανάγκες ε, αυξάνουν όταν μιλάμε για την καταπολέμηση της φτώχειας, το πρόγραμμα του 2020 κλπ. κλπ. Τώρα, στην ε, Περιφερειακή Επιτροπή ε, συζητήσαμε αν μπορούμε να ε, περιλάβουμε το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, το στρατηγικό πλαίσιο θέμα της ισότητας μεταξύ ανθρώπων και γυναικών και νομίζω ότι τούτο είναι μεγάλο βήμα όταν ομιλούμε για πολιτική συνοχής στα ευρωπαϊκά ταμεία. Είναι μια νέα προσέγγιση και όχι τόσο νέα. Δηλαδή όλο και περισσότερες επιτροπές και όχι μόνο οι συγητές κατανοούν το ζήτημα της ισότητας των φύλων και της ενσωμάτωσης στο βασικό κορμό. Και νομίζω ότι η κυρία Κράτσα όταν μίλησε για τις επενδύσεις στην Ευρώπη ορθώς επεσήμανε ε, ότι πρέπει να υπάρξουν δυνατότητες επιχειρηματικότητας για τις γυναίκες ιδιαίτερα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο. Ευχαριστώ και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Μπιλμπάου παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρο, ζητώ συγγνώμη που έφτασα με καθυστέρηση στην συνεδρίαση. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεση. Νομίζω είναι ένας τρόπος για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ισότητας με τρόπο εγκάρσιο και σε σχέση με τις τροπολογίες θεωρώ πως χρειάζεται να πάμε λίγο παρακάτω και να κάνουμε κάποιες ε, βελτιώσεις προτάσεις. Σε πολλές από αυτές ε, αναφέρουμε ότι τα προγράμματα θα πρέπει να εξαλείψουν τις διακρίσεις ανάμεσα σε άνθρωποι και γυναίκες αλλά δεν αναφέρονται σε κάποιες ε, προτάσεις ε, προκειμένου να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο θεωρούμε και ονομάζουμε ως θετική διάκριση. Εντάξει, στο Κοινοβούλιο έχουμε κάνει πάρα πολλές ε, δηλώσεις και διακηρύξεις, ανακοινώσεις σε γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις κλπ. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχουμε προχωρήσει ικανοποιητικά. Η έκθεση λοιπόν σε αυτή την κατάσταση κρίσης που αντιμετωπίζουμε ποινή. Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο, ξέρουμε ότι η ένδυα πλήττει περισσότερο τις γυναίκες ε, και ειδικά τα παιδιά. Εγώ ως ε, γενική παρατήρηση, μόνο ότι συμφωνώ με τις προτάσει, θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε λίγο παραπέρα και να ορίσουμε σε αυτόν τον κανονισμό πώς ε, επιθυμούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία ανάμεσα στι γυναίκε, αυτή η ισότητα μέσω των ταμείων. Και Συνοψίζοντας, ε, η ανάγκη πρόθεση ό,τι ανάμεσα στους άντρε και γυναίκε είναι, είναι μια σταθερή και υποφορά σε όλε τις τροπολογίε. Θα πρέπει να τονίσουμε πρώτον ότι οι στατιστικές ε, και οι πληροφορίε που υπάρχουν θα πρέπει να ε, θίξουν αυτό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει σαφής πληροφόρηση για να γνωρίζουμε αλλά και να υπολογίσουμε, να μετρήσουμε ποια είναι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση της εφαρμογής των ταμείων και αλλά όπως είπα ισότητα ναι, αλλά όταν μιλάμε για ταμεία θα πρέπει να πούμε πώς κρίνουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτή την ισότητα μέσω ταμείων. Οι επιχειρήσεις ε, που ιδρύονται από γυναίκες θα πρέπει να λαμβάνουν κάποια περαιτέρω βοήθεια. Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν ε, γυναίκες θα πρέπει να την κάνουν κάποιας περαιτέρω βοήθειας. Ε, αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε, διότι αντιθέτω, θεωρώ ότι θα παραμείνουμε μόνο σε επίπεδο δηλώσεων και εντάξει, καλά τα λόγια, αλλά θα πρέπει να εργαστούμε και να φέρουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και τέλος ε, θα δώσω το λόγο στον συγκίτρια κυρία Ζούμπερ, έχει το Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για την συμμετοχή τους στην συζήτηση. Φυσικά τώρα θα προχωρήσουμε με την αξιολόγηση των ε, τροπολογιών. Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε προτάσεις και συμβασμούς και είμαστε φυσικά διατεθειμένοι να πετύχουμε πρόοδο ομού για να υπάρξει περαιτέρω διευκρίνηση του κειμένου και να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα έπρεπε να περάσουμε στο σημείο 5, να πάμε πίσω, αλλά δυστυχώς αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, γιατί έχουμε μόνο 7 λεπτά μέχρι την έναξη των ψηφοφοριών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει το σημείο 5 να το περάσουμε για σήμερα το απόγευμα στις 15.00. Όχι, όχι, συγγνώμη μετά από την κοινή συνάντηση με την ε, Επιτροπή Ιουρί. Θα κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαλυματάκι, αλλά 10 και 30 ξεκινάμε τις ψηφοφορίες.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 Good morning, everybody. We will uh, now start. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, περνούμε τώρα στην διαδικασία της ψηφοφορίας και απλώς θα ήθελα τώρα να πάμε πίσω στο σημείο 6 γιατί ξέχασα να σας πω κάτι. Πρέπει να ανακοινώσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, καταληκτική ημερομηνία είναι 4 Ιουνίου, 5 η ώρα το απόγευμα και η Επιτροπή θα συζητήσει το θέμα στις 20 και 21 Ιουνίου και θα ψηφίσουμε στις 11 Ιουλίου. Αφού το ανακοίνωσα αυτό τώρα, περνούμε στο σημείο 7 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ησυχία παρακαλώ. You are... Όπως συνήθω λέω, είστε εξαιρετικά ελεύθεροι να ομιλείτε όσο περισσότερο θέλετε, αλλά έξω από αυτή την αίθουσα. Αυτό λέω συνήθως. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. το σημείο 7 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατάργηση του κανονισμού. Δεν υπάρχει συγητής και συνεπώς μπορούμε να αρχίσουμε την ψηφοφορία αμέσως. Θέλει κανείς να λάβει το λόγο? Όχι. Αρχίζουμε την ψηφοφορία λοιπόν. Τροπολογία υπαριθμών 2. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Πέρα στις ψηφοφορίες. πέρα απορρίπτεται λοιπόν πρέπει να κοιτάζετε τη μικρή οθόνη έτσι Περνούμε στην τροπολογία 18. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπερθμών 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνούμε στην τροπολογία υπαριθμών 20. Ξεχωριστή η ψηφοφορία σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία Α, να ελέγξουμε την 27 παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Δεν έχει καμία σημασία, είναι 16 με 10. Ξεκάθαρα εγκρίνεται. Θα πάω... Ναι, θα προχωρήσω πιο αργά. Τροπολογία 28. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε την 31 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Άζε το συγγνώμη λέει ο μηνυτής. Επαναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία υπαριθμών 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία. Νομίζω ότι ε, πρέπει να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα στην ε, εκπαίδευση. Μα, ε, με συγχωρείτε, πρέπει να περιμένουμε στατιστικά στοιχεία που θα αποδείξουν ότι τα στερεότυπα ε, ισχύουν. Είναι ασυμβίβαστα αυτά. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να ψηφίζουμε ό,τι να είναι. Δεν έχει κανένα νόημα. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη κυρία Λόλινγκ. Δεν κάνουμε συζήτηση τώρα. Είμαστε σε διαδικασία ψηφοφορίας. Διακόπτη η κυρία. Η γραμματεία πρέπει να μας πει ότι, να μας πει ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίζουμε έτσι ανόητα ο Πρόεδρος. Είμαστε τώρα στη διαδικασία της ψηφοφορία και εξαρτάται από εσά τα μέλη να αποφασίσετε αν αυτό είναι καλό ή κακό. Όχι, λέει η κυρία Λούλεγκ. Κοιτάξτε, υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες θα πρέπει να κριθούν ως απαράδεκτες, διότι ζητούν πράγματα που ε, δεν ισχύουν γιατί τα στατιστικά στοιχεία συγκαλύπτουν την πραγματικότητα. Μα πρέπει να περιμένουμε τα στατιστικά στοιχεία για να δούμε ότι υπάρχουν ε, στερεότυπα. Όχι, ο πρόεδρος διακόπτει. Κοιτάξτε, κάνετε συζήτηση τώρα. Όχι, δεν κάνω συζήτηση, λέει η κυρία Λόλου. Η γραμματεία στο μέλλον πρέπει να εξετάζει τις τροπολογίες αν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ή όχι. Ο πρόεδρος διακόπτει. Συνεχίζουμε και ψηφίζουμε την τροπολογία επαριθμών 32. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε τροπολογία υπαριθμών 32. The vote is closed. Πέρας της Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε ε, ε, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 11. It's adopted. It wasn't so clear from what I'm sitting. Λοιπόν, εγκρίνεται, είναι σαφέ. Άρα λοιπόν οι 1 και 10 καταπίπτουν και ψηφίζουμε την τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 Α, θέλετε να ελέγξουμε τη 14. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 14. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος και άρχεται η ψηφοφορία. Has everybody voted? Ψηφίσατε άπαντες. Όχι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε λοιπόν. Συγχαρητήρια στην συγγετρία. Τώρα περνούμε στο σημείο υπαριθμών 8. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την περίοδο 2014-2020. Τροπολογία υπαριθμών 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές δεν είναι αρκετά σαφές θα ελέγξουμε την 22 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία The vote is closed. It's adopted. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνούμε στην τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 7. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 12 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 14 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Το σύνολο του ψηφίσματος άρχεται η ψηφοφορία για ολόκληρο το κείμενο. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε το σχέδιο ψηφίσματος. person is there, you can. As good as they Okay. Okay, we then moving on to item number nine, establishing a European. Ε, τώρα στο 9, δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας. Ας αρχίσουμε αμέσως την ψηφοφορία για την τροπολογία 25. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ να σηκώσετε τα χέρια σας. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική λύση 1, Υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 4, ξεχωριστή ψηφοφορία, το πρώτο μέρος. Ψηφίζουμε το πρώτο μέρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 τώρα. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 36, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να το επαληθεύσουμε. Πάλι, τροπολογία 15, άρχιτη ψηφοφορία. Κλείνει. Απορρίπτεται η τροπολογία 15. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Συγχωρείτε. Θα, θα ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες 2 και 14. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 16, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ας υπαλληθεύσουμε το 17. Θα το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για το 17. Κλείνει. Όχι, με συγχωρείτε. Όχι, όχι, όχι. Ακυρώνεται. Όχι, δεν είναι. Έγινε κάποιο λάθος, θα μας για το 17. Τώρα αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 17. Τώρα. Κλείνει. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Ποιοι είναι υπέρ, είναι ξεχωριστή ψηφοφορία σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23, ποιοι υπέρ, κατά, αποχές. Λάθος έκανε ο πρόεδρος. Oh, sorry, sorry. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. Έκανα λάθος, λέει ο πρόεδρος. Ναι, έκανα λάθος. Μιλάμε για την τροπολογία 24, λάθος έκανα, με συγχωρείτε. Τροπολογία 24, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε όλο το ψήφισμα, αρχίζει η ψηφοφορία. sorry, yes, I had to check because I have, I, I had amendment 23 in my paper. Το δικό μου το χαρτί είχα μια τροπολογία 23, προφανώς δεν την είχατε εσείς. Γι' αυτό έκανα λάθος. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας. Yeah, sorry, it's adopted. Sorry. Εγκρίνεται, με συγχωρείτε, δεν το είπα ότι τελικά εγκρίνεται, φυσικά. We can Έρχομαι στο 10. Προπολογισμό 2013, εντολή για τον τριμερή διάλογο. Κύριε Χόνιμπολ, θέλετε να πείτε κάτι, ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις συζητητές. Ήταν ε, μια δύσκολη διαδικασία, αλλά καταλήξαμε σε μια συμβαστική λύση και είμαι ευγνώμων σε όλους για τη βοήθειά τους και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ερχόμαστε τώρα στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, καταπίπτει όχι. Η τροπολογία 3, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 4 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίθηκε. Ας το υπαλληθεύσουμε όμως. Τροπολογία 6 γίνεται επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία την τροπολογία 6. Κλείνει. Εγκρίνεται. Ναι, είναι σαφές, είναι σαφές. Τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, τώρα ερχόμαστε στη συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το οποίο σημαίνει ότι πάμε στη συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20. 20. Τροπολογία 20. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Έχει αποσυρθεί, συνεπώς ε, δεν θα την ψηφίσουμε. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατόπιν το 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. That means we 37. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, 39 καταπίπτει. Τώρα θα ψηφίσουμε τη 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. We're going to vote on amendment 44, yeah. We vote on amendment 44. Those... Τροπολογία 44. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι πρέπει να επαληθεύσουμε την ψηφοφορία εδώ. Τροπολογία 49, αρχίζουμε να ψηφίζουμε, κλείνει. Απορρίπτεται η 49. Τροπολογία 50, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω και εδώ πρέπει να κάνουμε μια επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 50. Ψηφίσατε. Κλείνει. Απορρίπτεται. The whole and the vote is now open. Αρχίζει η ψηφοφορία για το σύνολο. Κατά... The vote is closed. Κλείνει. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια Περνάμε στο σημείο 11. γιατί κάνουμε την πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα κλπ. Θα εξετάσουμε τις προφορικές τροπολογίες ομού και μετά θα περάσουμε στις φορές, όχι. Διαφωνείτε. Υπάρχουν ενστάσεις, όχι. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν επί του συνόλου. Όχι. Ψηφίζουμε την πρώτη τροπολογία και μετά θα ψηφίσουμε τις υπόλοιπες ομού, on Α, όχι, διαφωνείτε, εντάξει μία-μία χωριστά. Εντάξει. No problem. Τροπολογία 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ε, Περνάμε στο 12. Ενίσχυση της αλληλεγγύης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του ασύλου. Μπορούμε να ψηφίσουμε on block εδώ, όχι. Εντάξει. Ξεκινάμε με τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Item number 13, the support for the European Regional. Περνάμε στο 13, Συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Δυτικής Συνεργασίας. Σας ερωτώ, μπορούμε να ψηφίσουμε on block. Όχι. Τότε ξεκινάμε με την τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Δεν μπόρεσα να καταλάβω. Το αποτέλεσμα άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός. Τροπολογία 3. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. εποχές Δεκτή. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. εποχές Δεκτή. σημείο 14, ειδικέ διατάξεις ε, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης και το στόχο επενδύσεις ε, την ανάπτυξη και την απασχόληση και για την κατάργηση του κανονισμού 1080-2006. Περάσουμε σε εξέταση των τροπολογιών. Μία προς μία. Ήταν διαφορετικός τρόπος να πω αυτό που έλεγα πριν. Αν θέλετε να ψηφιστούν on block ή αν θέλετε να περάσουμε σε ψήφιση μία προς μία είπα να αλλάξω. Λοιπόν, τροπολογία 4, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Προπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Να περάσουμε στο σημείο 15, πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία. Μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Ξεκινάμε με την τροπολογία 4. Ψήφι Κατά. Αποχές. Δεκτή. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως πρέπει να παληθεύσουμε άρχιτη ψηφοφορία πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά εποχές. Ας επαληθεύσουμε. Τροπολογία 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τώρα στην τροπολογία 32 θα ψηφίσουμε μόνο την διαγραφή κλπ. Το υπόλοιπο καλύπτεται. Τροπολογία 32 λοιπόν υπέρ κατά αποχές. Θα επαληθεύσουμε άρχιτη ψηφοφορία επί της τροπολογίας 32. Έληξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 7 καταπίπτει, δεν ψηφίζεται, 7,5-33, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, εποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 10 υπέρ κατά Αποχές. δεκτή 35 κατά πίπτη 36 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή οι 11, 37 και 38 καταπίπτουν. Περνάμε στην τροπολογία 39. Ψήφι περ Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 12 καταπίπτει. Περνάμε στη 40. Ψήφι περ Κατά. Αποχές. Δεκτή. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 42 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 43 υπέρ κατά <clears throat> αποχές ας επαληθεύσουμε η τροπολογία 43 άρχεται η ψηφοφορία της ψηφοφορίας εγκρίθηκε Επαναλαμβάνουμε ψηφοφορία επί τη 43 μετά από αίτημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία εγκρίθηκε. Η 13 καταπίπτει. Περνάμε στην 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 20, τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε την 20 υπέρ. Ε, συγγνώμη, ηλεκτρονικά. Έληξη ψηφοφορία. Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Δεν ψηφίσατε πριν, δεν σηκώσατε χέρια σας. Τροπολογία 21, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 22, υπέρ. Κατά αποχές ας επαληθεύσουμε τροπολογία 22 ψηφίζουμε ηλεκτρονικός του ψηφοφορία πέρας απορρίφθηκε συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε στην 25 ψηφιπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή οι δύο καταπίπτει ψηφίζουμε την τρία. ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην εισηγητρία. Και πηγαίνουμε στο σημείο 16. Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια. Όπω είπα προηγουμένω, δεν θα ψηφίσουμε από αυτού. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων και η κυρία Γκόμε θα καταθέσει τι τροπολογίε τη συνολικά. Διότι θα έχετε τη δυνατότητα. Διότι έχετε τη είχατε τη δυνατότητα να τι δείτε προηγουμένω. Α, αλλά δεν είναι εδώ η κυρία Γκόμες. Δεν είναι εδώ η κυρία Γκόμες. Ρωτάω, υπάρχει κανένα άλλο που θα ήθελε να λάβει το λόγο σε αυτό το, θέ, στο σημείο αυτό. No. In that case we... Όχι, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να, να αφήσουμε προς το παρόν το 16 και έχουμε πολύ χρόνο για, το, για τις υπόλοιπες ε, ψηφοφορίες γιατί έχουμε στη διάθεσή μας 15 λεπτά μέχρι την κοινή συνεδρίαση και άρα μπορούμε να συζητήσουμε το σημείο 5. So then we go back to item 5 that we didn't have time Σημείο 5 λοιπόν. Έχουμε χρόνο να συζητήσουμε το σημείο 5 τώρα. Θα δώσω λοιπόν την Προεδρία στην κυρία Ρόκα. Ωραία. Με... Είναι μεγάλη τιμή που την αναλαμβάνω. Ιδιαίτερος, διότι ο συγγετής πέραν της ιδιότητάς του του Προέδρου αυτής της Επιτροπής κατόρθωσε να παραγάγει ένα εμπεριστατωμένο κείμενο. Πώς λοιπόν οι γυναίκες θα μπορέσουν να ενταχθούν στην μεγάλη αποστολή της ε, πράσινης οικονομίας. Κύριε Ισηγητά, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ, λέει ο και πρόεδρος. Θα ήθελα να αρχίσω αναφερόμενος καταρχήν πώς δούλεψα στο παρελθόν και πώς θα συνεχίσω να δουλεύω στο μέλλον και μετά θα ε, σχολιάσω το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω πολλά μέλη και πολιτικές, από πολλές πολιτικές ομάδες, διότι συμβάλλατε, συνεισφέρατε σημαντικά στην ε, σύνταξη της έκθεσης αυτής. Ε, προηγήθηκε μια διαδικασία διαβούλευσης όπου ε, μπόρεσα να λάβω υπόψη πολλές απόψεις και προτάσεις οι οποίες ήταν πολύ καλές και προσπάθησα να περιλάβω το μέγιστο δυνατό αριθμό αυτών. Δυστυχώς έχουμε περιορισμούς χώρου ως προς τον αριθμό των χαρακτήρων που μας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε σε μία έκθεση. Ε, έκανα το καλύτερο που μπορούσα για να περιλάβω όλες τις προτάσεις, αλλά δυστυχώς δεν χωρούσαν όλες. Γι' αυτό λοιπόν ε, εστιάστηκα σε αυτές που θεωρούσα ότι ήταν απολύτως απαραίτητες να περιληφθούν. Αλλά βεβαίως εσείς τα μέλη της Επιτροπής θα συμβάλλετε στη βελτίωση αυτής της έκθεσης και γι' αυτό περιμένω με ανυπομονησία να ακούσω και τις ε, τροπολογίες και με αυτόν τον τρόπο θα με βοηθήσετε ώστε να περιλάβω και αυτά που δεν κατόρθωσα να περιλάβω. Η έκθεση βασικά καλύπτει τρεις ιδέες, ισότητα, περιβάλλον και οικονομία. Τρία θέματα. Η δομή της έκθεσης εδράζεται σε κάποιες παραδοχές που αποτελούν και το πλαίσιο αυτών των προτάσεων. Ε, δίνουμε τον ορισμό της πράσινης οικονομίας, αλλά θέλουμε ταυτόχρονα της, ε, την αηφόρο οικονομία. Υπάρχει κεφάλαιο για τις μεταφορές, για πράσινες θέσεις εργασίας και ολοκληρώνεται η έκθεση με ένα κεφάλαιο για τις διεθνείς σχέσεις. Σημείο εκκίνησής μου στην έκθεση αυτή ήταν ότι οι μεταβολές οι οποίες επιτελούνται στο περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, οι διάφορες αλλαγές στα οικοσυστήματά μας συνδέονται άρρηκτα με τις συνθήκες διαβίωσής μας αλλά και με την ευημερία μας, την ευζωία μας. Μερικές φορές πιστεύουμε ότι μπορούμε να οικοδομούμε, να κατασκευάζουμε όσο πολύ όσα θέλουμε και όσο πολύ θέλουμε ή να καταναλώνουμε, να καταναλώνουμε όσο επιθυμούμε, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι, διότι αν καταναλώσουμε όλους τους πόρους του περιβάλλοντος, η κοινωνία δεν θα μπορέσει να επιβιώσει, δεν θα υπάρχει ευημερία. Ε, και συνεπώς δεν μπορούμε να περάσουμε και την όλη ευθύνη στις επόμενες ε, γενναίες. Δηλαδή να πούμε ας λύσουν οι επόμενες γενναίες τα ζητήματα αυτά. Πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα. Άρα λοιπόν ένα από τα σημεία κίνησής μου είναι ότι χρειαζόμαστε μια πράσινη οικονομία. Αλλά ο ορισμός μου της πράσινης οικονομίας δεν αφορά μόνο να πούμε στους ανεμόμυλους, στους ε, ε, στα ελληνικά πάρκα κλπ. κλπ. Αυτό που εννοώ εγώ με, την πράσινη, με τον όρο πράσινη οικονομία είναι μια κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμη και αηφόρο οικονομία σε όλες τις, τις πτυχές. Τι σημαίνει όμως κοινωνική αηφορία. Εκεί επισέρχεται η κοινωνική δικαιοσύνη στο ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και μεταξύ ανθρώπων και γυναικών, διότι η κοινωνική διάσταση είναι εξίσου σημαντική με την πράσινη οικονομία όπως ας πούμε το, η ισορροπία των οικοσυστημάτων. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με την περιβαλλοντική πτυχή χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την κοινωνική διάσταση. Διότι υπάρχει τεράστια κοινωνική αδικία στον κόσμο και υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έτσι βλέπω εγώ την έννοια πράσινη οικονομία. Ένα άλλο σημείο εκκίνησης. Η ρόλη είναι η ρόλη των φίλων άνδρες και γυναίκες έχουν διαφορές ως προς την επιρροή του στο περιβάλλον, ως προς τα εισοδήματα, ως προς τον βαθμό εξουσίας κλπ. Και επίσης τα σχήματα και οι συνήθειες κατανάλωσης είναι διαφορετικές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Άρα λοιπόν άνδρες και γυναίκες επηρεάζουν το περιβάλλον κατά διαφορετικούς τρόπους. Οι άνδρες χρησιμοποιούν περισσότερα ιδιωτικά, οι γυναίκες δημόσιες μεταφορές, κάτι το οποίο επηρεάζει σε τεράστιο βαθμό το περιβάλλον. Οι γυναίκες είναι περισσότερο vegetarians. Πώς... Οι γυναίκες λοιπόν είναι περισσότερο χορτοφάγια από τους άνδρες. Όλα αυτά επηρεάζουν το περιβάλλον. Ένα θέμα το οποίο εμφανίζεται συχνά σε αυτή την Επιτροπή είναι το θέμα των στατιστικών. Αν δεν υπάρξουν δείκτες, δείκτες για τα δύο φύλλα, τότε είναι δύσκολο να κάνει κανείς προτάσεις για λύσεις. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία, κατανομή, κατά των στατιστικών στοιχείων. Και προσπάθησα κάνοντας αυτή τη δουλειά, αναζήτησα αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο να βρει κανείς αυτά τα στοιχεία. Δεν μπορεί κανείς να βρει στατιστικά στοιχεία με βάση την κατανομή κατά φύλλο. Ένα άλλο σημείο είναι ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες λήψης αποφάσεων στο στους κόλπους της οικονομίας και στο πλαίσιο μιας πράσινης οικονομίας. Δηλαδή η πολιτική λήψη αποφάσεων δεν είναι 50-50, ούτε καν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι γυναίκες πρέπει να εμπλακούν σε σοβαρές αποφάσεις στο οικονομικό τομέα και πρέπει να υπάρξει αυτή η εμπλοκή κατά ισότιμο τρόπο για το τι δρόμο θα πάρει η οικονομία στο μέλλον και στις δια... δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις και στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές. Λίγες είναι οι γυναίκες που εμπλέκονται. Πρέπει όμως οι εμπειρίες των γυναικών να ληφθούν υπόψη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Χωρίς αυτό δεν λαμβάνουμε υπόψη την εμπειρία και την άποψη του μισού του πληθυσμού της γης. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε και το τοπικό επίπεδο όπου θα πρέπει να εμπλακούν οι γυναίκες. Υπάρχει ένα θέμα για τις αναθρωπιτισόμενες χώρες. Ε, οι μελέτες και η έρευνα δείχνουν ότι αν εκπαιδεύσει κανείς τις γυναίκες μπορεί να προλάβει καταστροφές, να προστατεύσει τα δάση, να συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας κλπ. Άρα το να δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες για να ασχοληθούν στην τοπική κοινωνία, το να δίνουμε περισσότερες εξουσίες στις γυναίκες έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Αυτά είναι τα σημεία εκκίνησης της έκθεσής μου. Αλλά τώρα να πω και δύο λόγια ως προς τις απαιτήσει. Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές ιδέες. Πρώτον, Πρέπει να θυμόμαστε ότι η οικολογική βιωσιμότητα θα πρέπει να προχωρήσει χέρι με χέρι με την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική αηφορία. Και τούτο σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, για τα οικοσυστήματα, την κατανάλωση, την ε, διατροφή, την ανάπτυξη, τις μεταφορές, την ενέργεια και τον ε, τομέα της... ευημερίας. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη αυτής της προοπτικής στο έγγραφο της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε για το 2020. Δεν υπάρχει καθόλου η προοπτική των φίλων σε αυτό το έγγραφο. Τώρα, τι σημαίνει ε, βιώσιμη κατανάλωση ή αηφόρος κατανάλωση, sustainable ε, consumption. Ε, να δούμε τι συζητάμε στις χώρες μας αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Θέλουμε όλη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έχει γίνει μια μορφή θρησκείας. Ε, θεωρείται κάτι απολύτως θετικό, όπως είναι η δημοκρατία και η ελευθερία, η ανάπτυξη. Καλά. Σαν να είναι, ας πούμε, ο χρυσός, η ανακάλυψη του χρυσού, η ανάπτυξη. Και αυτό είναι επίσης πρόβλημα. Τι σημαίνει ανάπτυξη? Σημαίνει ότι παράγουμε περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι καταναλώνουμε περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες. Σημαίνει ότι δημιουργούμε όλο και περισσότερα για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των ατόμων. Ας πούμε, ικανοποιούμε την ανάγκη της τροφής, της καλής ζωής, των ταξιδίων κλπ. Δηλαδή δεν έχει νόημα να παράγουμε πράγματα έτσι για να τα παράγουμε και δεν μπορεί να μετατρέπεται η ανάπτυξη σε μορφή θρησκείας. Αν κανείς κοιτάξει το ΑΕΠ, ασφαλώς, αυτό είναι ένα μέτρο της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά πρέπει κανείς να λάβει υπόψη και άλλους δείκτες, ας πούμε, η κοινωνική ευημερία, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτά δεν αντανακλώνται στο ΑΕΠ και βεβαίως αν κανείς ας πούμε ρίξει πετρέλαιο στη θάλασσα και μετά ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού αυτό μπορεί θαυμάσια να συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ αλλά είναι καλό αυτό πρέπει δηλαδή να βρούμε δείκτες οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη και άλλες πτυχές ε, επίτευξη δηλαδή των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων θα πρέπει να είναι ένας δείκτης παραδείγματο χάρη το ΑΕΠΤ παραδείγματο χάρη δεν αντανακλά καθόλου το έργο των γυναικών στα σπίτια, αυτό που κάνουν οι γυναίκες στο σπίτι τους. Πρέπει να λάβει υπόψη την κοινωνική δικαιοσύνη, το περιβάλλον και την ισότητα. Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνουν ότι η οικονομική πολιτική των χωρών μελών πρέπει να τροποποιηθεί αν θέλουμε να επιτύχουμε την πράσινη οικονομία, διότι πρέπει να εστιάσουμε στην κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Θα πρέπει δηλαδή να αποφύγουμε τη συνέχιση των βλαπτικών για περιβάλλον δραστηριοτήτων. Ολόκληρη η κατανάλωση περιλαμβανομένη των, και των τροφών θα πρέπει να γίνουν στα, στο πλαίσιο ορίων. Εδώ δηλαδή στη Δύση, ας πάρουμε τη δική μου χώρα, τη Σουηδία, αν ο καθένας προσπαθούσε να ζήσει όπως εμείς ζούμε, τότε θα χρειαζόμασταν 3,5 πλανήτες. Δυστυχώς δεν έχουμε τρεις πλανήτες, έχουμε μόνο έναν πλανήτη. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε πολύ προσεκτική σχήση των πόρων μας. Υπάρχουν φτωχοί και στη δική μας χώρα και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αυτοί χρειάζονται αυξημένη κατανάλωση και ανάπτυξη. Άρα πρέπει να διασφαλίσουμε κάποια προοπτική ισότητας. όχι μόνο στη δική μας δουλειά, αλλά και σε όλες τις πτυχές της χάραξης πολιτικής. Ένα άλλο κεφάλαιο είναι οι βιώσιμες μεταφορές. Γιατί, Γιατί οι μεταφορές είναι απαραίτητες και για τους άνδρες και για τις γυναίκες, για τα ταξίδια και για την επικοινωνία υπάρχει η περιβαλλοντική πτυχή, αλλά υπάρχει και το σκέλος το κοινωνικό, διότι είναι θέμα κινητικότητας και ελευθερίας οι μεταφορές. Άρα λοιπόν, κοινωνικός σχεδιασμός, σχεδιασμός ε, κίνησης, πρέπει να εστιάσει και στον περιορισμό, στη μείωση της κίνησης. Ξέρουμε ότι οι άνδρες χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Γι' αυτό και οι επενδύσεις σε αυτοκινητοδρόμους είναι πολύ περισσότερες από ό,τι ας πούμε στα δημόσια μέσα μεταφοράς. Τώρα, στην ψηφιακή εποχή, αν έχει κανείς ένα καλό σχεδιασμό, τότε δεν χρειάζεται να αυξήσει τα αστικά δίκτυα. Μπορεί να έχει πολύ πιο αποτελεσματικές ε, υπηρεσίες μεταφορών. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να αγοράζουν αυτοκίνητα και ε, τώρα όλο και περισσότερο οι γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητα όσο και οι άνδρες. Και τις επιπτώσεις αυτού του φαινομένου πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Χρειαζόμαστε επίσης μια ιεραρχία μεταφορών όπως υπάρχει η ιεραρχία αποβλήτων. Αν κοιτάξουμε πώς ταξιδεύουμε, θα πρέπει να δούμε ε, πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Α, χρησιμοποιώντας τα ε, ψηφιακά μέσα θα μπορούσαμε να περιορίσουμε τα ταξίδια. Ε, Πρώτο λοιπόν, περιορισμός ε, της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου, δεύτερο δημόσιες μεταφορές ε, και μόνο τελευταία, τελευταία επιλογή ε, να ταξιδεύει κανείς με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο. Εντάξει, αν με προσκαλέσουν να πάω στην Αυστραλία σε ένα συνέδριο, αναγκαστικά δεν θα πάρω το ποδήλατό μου, αλλά θα κάνω κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πράσινες θέσεις εργασίας, πράσινη απασχόληση είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Τι, προσπαθώ να διευρύνω τον όρο της πράσινης οικονομίας για να περιλάβει περισσότερα από όσα αρχικά προβλέπονταν. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τούτο αφορά στην ενέργεια, τις κατασκευές, τα αποβλη, διαχείριση αποβλήτων κλπ. Όλους αυτούς τους τομείς. Υπάρχουν βεβαίως πράσινες θέσεις απασχόλησης και στον τομέα των υπηρεσιών υπάρχουν θέσεις απασχόλησης στα σχολεία, στην ε, ε, ε, ιατρική φροντίδα, υπάρχουν πράσινες θέσεις απασχόλησης και για άνδρες και για γυναίκες. Και θα πρέπει άνδρες και γυναίκες να έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας πρέπει να λάβουμε υπόψη την τρέχουσα αγορά εργασίας για να διαμορφώσουμε και τη μελλοντική πράσινη αγορά εργασίας. Άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να δουλέψουν σε κλάδους της πράσινης τεχνολογίας, όπου κυριαρχούν οι άνδρες. Χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη κατάρτιση και χρειαζόμαστε και ε, κατάρριψη των ε, στερεοτύπων φίλου, ως προς το φίλο. Ασφαλώς πρέπει περισσότερες γυναίκες να δουλέψουν στους πράσινους τομείς, αλλά επίσης και περισσότεροι άνδρες να δουλέψουν στο... Internationella relationer så tror jag att e ε, περισσότεροι άνδρες λοιπόν να δουλέψουν στο, στον τομέα των κοινωνικών παροχών, κοινωνικών υπηρεσιών. Ε, Επίση πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι εξελίξει τη αναπτυσσόμενη χώρε. Χρειαζόμαστε καταρχήν οικονομικού δείκτε πέραν του ΑΕΠ δηλαδή δείκτες που θα μετρούν τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να μετρούμε την αποτελεσματικότητα προγραμμάτων στην, στην ισότητα των δύο φύλων. Αν μπορέσουμε και μετρήσουμε αυτό το στοιχείο, δηλαδή την επίδραση στην ισότητα των φύλων, τότε θα μπορούσαμε ας πούμε να βρούμε ε, τι μπορεί να γίνει ας πούμε για την ενέργεια ή το καθαρό νερό. Το καθαρό νερό είναι καθοριστική σημασία για τις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό το χρειάζονται οι γυναίκες, οι γυναίκε για το σπίτι και τείνουν αυτές να έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν νερό για την οικογένεια και μάλιστα καθαρό νερό. Αυτό συνδέεται άμεσα με τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Μπορεί αυτό να αναπτυχθεί σε τοπικό επίπεδο. Πολλέ οικογένειε χρησιμοποιούν ε, χρησιμοποιούν ας πούμε κάποιο καύσιμο για να μαγειρέψουν το φαγητό. Αλλά αν κανείς έχει ένα ε, ηλιακό, μια ηλιακή συσκευή θα μπορούσε να αποφύγει τις ε, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία από την χρήση ενός καυσίμου μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη καθώς θα αναπτύσσουμε τα νέα μας προγράμματα ενώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη γνώση και την εμπειρία των αυτοχθόνων πληθυσμών. Ε, υπάρχουν ήδη λύσεις που έχουν δοθεί από παλιά. Οι τοπικοί πληθυσμοί έχουν τεράστια βάση γνώσεων, ιδιαίτερα οι γυναίκες και πρέπει εμείς να κάνουμε βέλτιστη χρήση αυτής της γνώσης. Επίσης, πρέπει τα προγράμματα και τα project της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να στοχεύουν και στην καταπολέμηση των ε, διακρίσεων μεταξύ των δύο ε, φύλων. Ας πούμε τα μικροδάνεια, μικρή έκταση δάνεια κλπ. που μπορούν να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών. Ε, χρειαζόμαστε συστήματα για τα φάρμακα. Να μπορούν οι φτωχές χώρες, οι αναπτυσσόμενες χώρες να παράγουν φθηνά φάρμακα. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό με την αιωλική ενέργεια, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν τέσσερι εταιρείε αυτή τη στιγμή που έχουν τις πατέντες για την αιωλική τεχνολογία σε ολόκληρο το κόσμο. Αλλά αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την μορφή ενέργειας ως μια βιώσιμη πηγή, δεν είναι δυνατόν να χρειάζεται κανείς να χρησιμοποιήσει τεχνολογία προ 15 ετίας ενώ υπάρχουν σύγχρονες πατέντες με μοντέρνα μέσα αλλά τις κρατούν στα χέρια τους δύο-τρεις εταιρείε. Άρα λοιπόν η... η ευημερία και το περιβάλλον κινδυνεύουν και χρειαζόμαστε μια πράσινη οικονομία η οποία θα είναι αηφόρος κοινωνικά αλλά και περιβαλλοντικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη ε, εκ μέρους Επιτροπής της Κομισιόν η, συνάδελφος ήταν εδώ για να εκπροσωπήσει την Επιτροπή. Αλλά επειδή έγινε κάποια αλλαγή της σημερινής διάταξης, νόμιζε ότι πρόκειτο να παρουσιαστεί στις το θέμα και γι' αυτό δεν μπόρεσε να είναι παρούσα. Γι' αυτό εμείς εμείς θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποια είναι η άποψη της Επιτροπής της Κομισιόν. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ζητώ συγγνώμη για την κυρία Μπάρμπαρα Μέρες και όλη συγκήτρια για αυτή την έκθεση. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα εδώ και μου ζήτησε να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της και έχει και ένα μικρό σημείωμα το οποίο ετοίμασε. Θα ήθε... Το σημείωμά είναι το εξή. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο της Επιτροπή, τον κύριο Γκούσταυσον, για την σύνταξη της έκθεσης για τις γυναίκε και την πράσινη οικονομία και ε, τη διακριτική μεταχείριση την οποία δυστυχώ αντιμετωπίζουν ακόμα οι γυναίκε για την πρόσβαση στην αγορά εργασία. Τη στιγμή που η πράσινη οικονομία αναπτύσσεται, η συμβολή των γυναικών είναι πολύ σημαντική σήμερα, επειδή σε όλου του τομεί οικονομία δραστηριοποιούνται οι γυναίκε και φροντίζουν την οικογένειά του παράλληλα αλλά συμβάλλουν και στις δομές της κοινωνίας τους αλλά και στις επιχειρήσεις οι ικανότητες και η συμβολή των γυναικών δεν αναγνωρίζονται παρκώ. Νέες ευκαιρίες της πράσινης οικονομίας θα πρέπει να επιτρέψουν να γίνουν τομεακές αλλαγές με νέες θέσεις εργασίας αλλά και με απώλεια θέσεων εργασίας. Ε, πρέπει να είναι πιο παρούσες οι γυναίκες σε τομείς όπου είναι μόνο οι άντρες παρόντες. Θα πρέπει να δούμε πώς η πράσινη απασχόληση ε, θα έχει χώρο για τις γυναίκες, μίσο που υπάρχουν μόνο άνδρες. Συνήθως οι γυναίκες δεν αμείβονται όσο οι άνδρες και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να επιτρέψουν να γίνει αυτή η αλλαγή προστατεύοντας τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, φροντίζοντας ε, προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν θέση απασχόληση στα υψηλά επίπεδα χρειάζεται μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τη θέση των γυναικών στην πράσινη οικονομία. Ε, επιθυμούμε να μην υπάρχει άνηση κατανομή μεταξύ εξειδικευμένων και μη εξειδικευμένων για να υπάρχει ποιοτική εργασία σε όλες τις θέσεις στην πράσινη οικονομία. Για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής μισθός και πρόσβαση σε αυτές τις θέσεις τις γυναίκες. Ε, η επαρκής κατάρτιση θα επιτρέψει στις γυναίκες να βρουν ε, θέσεις, σε θέσεις διοίκησης στην πράσινη οικονομία και θα τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε βιώσιμες τεχνολογίες στον τομέα της ε, διοίκησης των μεταφορών, τα μέσα ενημέρωσης, τις επικοινωνίες, ώστε οι γυναίκες να συμμετέχουν περισσότερο ε, σε βιώσιμες εργασίες. Θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη συμμετοχή ε, στο επίπεδο λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων θα πρέπει να υπάρχουν γυναίκες, στα πάνελ εμπειρογνωμόνων ε, της πράσινης οικονομίας. Επίσης, ίση συμμετοχή στα όργανα λήψης αποφάσεων για να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και επιθυμίες των γυναικών. Είναι ουσιαστικό να ενσωματωθεί αυτό το σκέλος του γυναικείου στην πράσινη οικονομία. Αυτό υπόθηκε και στον ΟΗΕ, διότι ε, χιλιάδες άτομα στις αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτώνται από βιομάζα και συχνά είναι οι γυναίκες που είναι υπεύθυνε να συλλέγουν αυτά τα προϊόντα που βγαίνουν από τη βιομάζα. Για παράδειγμα, τα κατάλοιπα της γεωργίας ή του ξύλου. Επίσης πρέπει να γίνουν επενδύσεις στις ε, λιγότερο ε, ρηπογόνα προϊόντα, στις ε, λιγότερο ρηπογόνες τεχνολογίες και θα πρέπει να υπάρχει κατάρτιση να δώσουμε αυτοπεποίθηση στις γυναίκες για να ξεκινήσουν μόνες τους επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ποιε θα είναι οι θετικές επιπτώσεις για τη γυναίκα, ώστε το καθεστώς της γυναίκας να βελτιωθεί. Ε, εκεί όπου δεν υπάρχει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να υπάρχουν ανάσχομες πηγές ενέργειας ώστε όλες οι περιοχές ε, να έχουν ενεργειακές πηγές ε, για να αξιοποιηθούν τοπικές εργασίες για τις γυναίκες. Καταλήγοντας, έχω πιστεί ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το σκέλος της ισότητας των φύλων στην πράσινη οικονομία και θα πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα για να βελτιωθεί η πρόσβαση των γυναικών στις ευκαιρίες που υπάρχουν στην πράσινη οικονομία θα λάβω υπόψη τις τροπολογίες ε, που αναφέρουν προγράμματα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, προκειμένου ε, οι γυναίκες να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις ευκαιρίες δουλειάς που γίνονται από την πράσινη οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το σημείο με αυτό το οποίο μας διαβάσατε. Καλά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για ε, την εργασία που μας παρουσιάσετε σήμερα το πρωί και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας πω από εκβάθους βάθους ότι θεωρώ ενδιαφέρον το γεγονός ότι επιμείνατε ότι για σας η πράσινη οικονομία δεν είναι μόνο η περιβαλλοντική οικονομία υπό τη στενή έννοια της λέξης. Και τονίσατε μάλιστα την κοινωνική βιωσιμότητα. Και νομίζω ότι εάν σε αυτό το τομέα κάτι πρέπει να κάνουμε είναι να μην περιοριζόμαστε μόνον στην πράσινη οικονομία, αλλά να τη συνδέσουμε με την κοινωνική βιωσιμότητα. Μας ε, δείξατε τον ενθουσιασμό σας και το όραμά σας Νομίζω ότι πρέπει πολλά να κάνουμε μαζί για να υπάρξει αυτό το άνοιγμα όσον αφορά την κοινωνική βιωσιμότητα. Και νομίζω ότι ο αγώνας θα είναι δύσκολος. Δεύτερο, τονίσατε την ανάγκη να υπάρχουν γενικές στατιστικές κατατομής. Βεβαίω μας χρειάζονται στατιστικές ανατομής, διότι πρέπει να αποδείξουμε τις ανισότητες που ορισμένοι δεν θέλουν να βλέπουν. Και συνεπώς θα πρέπει επίσης να δραστηριοποιηθούμε, να κινητοποιηθούμε. Αυτό θα είναι ο δεύτερος αγώνας που θα πρέπει ε, να κάνουμε μαζί για να έχουμε αναλυτικές στατιστικές που θα αποδείξουν ότι υπάρχουν κοινωνικές δυσλειτουργίες και ποιες είναι οι εξελίξεις που επιθυμούμε. Το τρίτο σημείο επί του οποίου συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, είναι η ισότητα στο επίπεδο λήψης αποφάσεων όλων των επίπεδων. Δεν μπορούμε να εξελιχθούμε σε αυτό το τομέα ούτε στα, στους άλλους τομείς εάν δεν υπάρχει αυτή η βούληση ισότητας στα ανώτατα επίπεδα των λήψεων αποφάσεων. Και αργότερα θα σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα γιατί τα πράγματα δεν πάνε πάντοτε πολύ καλά. Δηλαδή, οι γυναίκε εκπροσωπούν το 50% του πληθυσμού και όλες οι χώρες μας επενδύουν πολύ για ισότητα κατάρτιση εκπαίδευση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και τελικά, τι γίνεται μετά. Υπάρχει μία λάθος μεταφορά αυτής της θαυμάσιας κατάρτισης των γυναικών, γιατί ακριβώς οι γυναίκες δεν βρίσκονται στα αξιώματα που αξίζουν, δεν ακολουθούν καριέρα την οποία τους αξίζει, δεν ανεβαίνουν αρκετά και δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Και τελικά αυτή η ανισομέρεια, αυτή η ανισότητα συνεχίζεται και διευρύνεται. Είπατε ότι ένα από τα μέσα για να καταπολεμήσει κανείς αυτή την ανισότητα, την ανισομέρεια, είναι σε τοπικό επίπεδο να αποτραπούν αυτές οι ανισομέρειες επιτρέποντας στις γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε θέσεις υπευθυνότητας. Εγώ ε, προέρχομαι από μια χώρα όπου η ισότητα είναι όχι μόνο νόμιμη αλλά και υποχρεωτική όσον αφορά τις τοπικές αρμοδιότητες και ευθύνε. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξή. Ας προσέξουμε, να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι οι γυναίκες περιορίζονται σε ευθύνες που αντιστοιχούν ε, σε γυναικεία πρότυπα, δηλαδή ο κοινωνικός τομέας, ο εκπαιδευτικός τομέας κτλ. Ενώ για να υπάρχει αυτή η κοινωνική βιωσιμότητα, οι γυναίκες πρέπει να έχουν ας πούμε, την Προεδρία τη επιτροπή των Δημοσιονομικών, ε, τη οικονομική επιτροπή, Επιτροπής, ενός Δημαρχείου, ε, μιας κοινότητας. Δηλαδή να δούμε τι επιπτώσει που έχει αυτό το θέμα της αρμοδιότητας υπευθυνότητα των γυναικών. Δηλαδή να δούμε όχι μόνο την ισότητα, αλλά και στην πραγματικότητα τι συμβαίνει και πού βρίσκονται οι γυναίκε στα ανώτατα κλιμάκια. Το δεύτερο σημαντικό σημείο, επί του οποίου ήθελα να μιλήσω, είναι η ανάπτυξη. Νομίζω ότι είπατε ότι πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη, συμφωνώ απόλυτα και είμαι πεπισμένη για το εξή. Ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια καμπή και τα κοινωνικά ζητήματα θα προσλάβουν πολύ μεγάλη σημασία, διότι η κρίση θα οδηγήσει σε κοινωνικές εξεγέρσεις και δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη το κοινωνικό σημείο, το κοινωνικό, κοινωνικός κρίκος, αυτή την αλυσίδα της κρίσης. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι σε αυτό το τομέα επίσης η θέση μας είναι και στρατηγική και πολιτική. Θα πρέπει να καλύψουν ένα χώρο εδώ. Και γι' αυτό το λόγο, στα πλαίσια αυτής της πράσινης οικονομίας, το κοινωνικό σκέλος θα πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να επιμείνω στο εξής. Οι γυναίκες αναλύουν διαφορετικά τα πράγματα και ε, όσον αφορά ε, η, την αλληλεγγύη και την αντιμετώπιση της σπατάλης, ε, οι γυναίκες μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η σπατάλη των τροφίμων, για παράδειγμα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ακόμα μερικά σημεία. Πρώτα απ' όλα, το θέμα των μεταφορών. Στην μελέτη σας αναφέρεται ότι ορισμένες κοινότητες ε, ίδρυσαν γραφεία χρόνου για να ληφθεί υπόψη αυτή η απόσταση μεταξύ ε, ανδρών και γυναικών που υπάρχει ακόμα. Θα ήθελα να σας πω να είσαστε προσεκτικοί. Προσοχή. Γιατί. Ε, επειδή αυτά τα γραφεία χρόνου έχουν πολιτικό χαρακτήρα και δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικά τις, τα, την πραγματικότητα. Και τώρα είναι κάτι το οποίο έχει λησμονηθεί. Απλά και μόνο αυτό ήταν μια δήλωση και μετά δεν έγινε τίποτα. Εγώ κατοικώ σε μια πόλη όπου υπάρχουν ε, διαμερίσματα με πολλά γραφεία χρόνου, όπως τα λέμε. Και πρέπει να σας πω ότι ε, δεν είχαμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, διότι αφού εξαγγέλθηκε αυτό το μέτρο, είχαμε αφήσει, το ξεχάσανε εντελώς. Και η πολιτική βούληση χρειάζεται για να συνεχίσουμε αυτό το στόχο, αν θέλουμε να έχει αποτελέσματα. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα τελευταίο σημείο, δηλαδή η καταπολέμηση των στερεοτύπων και ε, αυτό σε όλα τα επαγγέλματα. το, το να γίνουν να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες σε ένα τομέα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όταν υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες σε ένα επάγγελμα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια υποβάθμιση του επαγγέλματος. Λοιπόν, ανάμεσα σε στερεότυπα, παρά το γεγονός ότι ορισμένα επαγγέλματα είναι πιο γυναικεία, ενώ άλλα επαγγέλματα δεν είναι θελκτικά για τις γυναίκες. Την προηγούμενη εβδομάδα στη δική μου την περιφέρεια επισκέφθηκα ένα χώρο όπου γίνεται κατάρτιση ε, συντηρητών ε, αιωλιακών ε, αιωλικών πάρκων που είχαν χρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Και ρώτησα πόσες γυναίκες είναι εδώ, βεβαίως, ήδη το ερώτημά μου ήταν μια φάδια και υπήρχε μόνο μια κοπέλα, μια γυναίκα. Ζήτησα πάλι πώς βρήκε δουλειά αυτή η κοπέλα στο τέλος της κατάρτισής της. Και ήταν η υπεύθυνοι της κατάρτισης, οι δάσκαλοι, καθηγητές μου είπαν όλος ο κόσμος την ήθελε, όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις ήθελαν να προσλάβουν αυτό το κορίτσι. Και είπα, ναι, θα, θα ξανάρθω εδώ για να δω στα επόμενα χρόνια πόσες γυναίκες θα έχετε. Λίγεται λοιπόν λόγος για αυτό το θέμα στην πράσινη οικονομία. Πρέπει κανείς να κάνει επισκέψεις επί τόπου και να, γιατί αν δεν ασκηθεί μεγάλη πολιτική πίεση νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Και τώρα η ε, κυρία τη νέο μέλος της Επιτροπής μας από τη Ρουμανία. Ευχαριστώ. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα είπατε, διότι η έκθεση αναλύει με τρόπο ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μένα τουλάχιστον κάποιες διαφορετικές θέσεις και απόψεις τις οποίες δεν είχα ακόμα σκεφτεί. Για μένα λοιπόν πρόκειται για μια νέα και καινοτόμα αντίληψη. Θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα. Ο Ιγαλίδας συνάδελφος μίλησε για την δυσκολία, για την σημασία της συμμετοχής των γυναικών στην διαδικασία λήψη αποφάσεων, όπου η Γαλλία είναι, θα έλεγα, πρωταθλητής αναφέρομαι στα περιφερειακά συμβούλια, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει διόλου στη Ρουμανία. Λοιπόν, η συνάδελφοι δεν είναι πάντα ικανοποιημένη, αυτό σημαίνει πως πολλά απομένουν να γίνουν και στη Γαλλία. Αλλά ίσως χρειαστεί να τονίσουμε το ότι πρέπει να συμμετέχουν γυναίκες σε όλα τα επίπεδα λήψης απόφασης και χάραξης πολιτικής. Και θα ήθελα να προτείνω το εξής όλα τα μέτρα τα οποία προτείνεται είναι βράχη μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, αλλά σε ό,τι φορά το ζήτημα θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις και υπολογισμοί μακροπρόθεσμοι ναι. και εδώ μπαίνουμε στον τομέα της εκπαίδευσης, ε, της κατάρτισης και εδώ οι γυναίκες έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Στην εκπαίδευση όμως, εκεί όπου οι γυναίκες έχουν την πλειοψηφία, η μισθή είναι πολύ χαμηλότερη, πολύ χαμηλή. Άρα κάτι θα πρέπει να γίνει ώστε οι δασκάλες ε, να ασχοληθούν ιδιαίτερα με τον τομέα της αηφόρου ανάπτυξης από την πιο τρυφερή ηλικία διότι τα παιδιά μας θα πρέπει να γνωρίζουν από μικρά ότι θα πρέπει να σέβονται τον, τη φύση, να τρέφονται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία θα πρέπει να τύχουν υπογράμμισης στην έκθεσή σας και να τονίσετε το ρόλο της γυναίκας ως μητέρα πρώτον αλλά και ως δασκάλα όπου τα παιδιά μας οι μελλοντικοί ενήλικες θα πρέπει να εκπαιδευτούν σωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τριβέτη. Επιτρέψτε μου να μίλησω κι εγώ και να σας, να επενέσω την προσέγγιση σας. Ξέρουμε ότι είσαστε επαγγελματικά αναμειγμένος στο ζήτημα της πράξης οικονομίας. Έχετε πολλά να μας πείτε. Και ε, αυτό το οποίο ξετίμησε ιδιαίτερα στο κείμενό σας είναι ότι μιλάτε για μηχανισμούς μείωσης της ένδυας ε, μέσω της πράσινης οικονομίας συνειδητοποιούμε ότι πολλοί από τους φτωχούς είναι φτωχοί διότι ε, στο παρελθόν πριν ότι κατά τη διάρκεια μάλλον της ε, κομμουνιστικής μας περίοδου ε, όλοι είχαμε δουλειά, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει τώρα. Τώρα λοιπόν βλέποντας ότι και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει ε, μεγαλώσει η ανεργία θα πρέπει να εξετάσουμε καλύτερο θέμα της πράσινης οικονομίας. Τώρα, οι νέοι δείκτες ε, εκτός από το ΑΕΠ είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Και θα θέλαμε να εργαστούμε πάνω σε αυτούς τους νέους δείκτες. Η κυρία Τριβέτη εφιώς είπε πως θα μιλάμε για πράσινη οικονομία και γυναίκες προσπαθούμε να προωθήσουμε το Think Green για την επόμενες γενιές αλλά και το ζήτημα της συνειδητοποίησης θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο. Θεωρώ λοιπόν ότι η απόψη σας περί green thinking ε, θα μπορεί να τύχει ιδιαίτερη προσοχής από τις γυναίκες ε, για να το προωθήσουν όπως είπα και εσείς, από, όπως υπόθηκε μάλλον νωρίτερα από την τρυφερή ηλικία. Εγώ φροντίζω μέσω του διαδικτύου να ενημερώνουμε συνεχώς για αυτά τα ζητήματα πώς ε, θα πρέπει να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, ειδικά οι γυναίκες που έρχονται από την ε, Ανατολική Ευρώπη, δεν έχουν αυτή την αντίληψη του Think Green. Εσείς ε, ως Βόρειος, ως Σουηδός, φυσικά επηρεάζεται τις δυνατότητες ε, που έχουμε και συμφωνούμε ότι οι γυναίκες έχουν πολλά να κάνουν. Κάτι ακόμα. Η υπεύθυνη για τη χάραξη πολιτική θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι έφτασε η ώρα να συμμετέχουν και οι γυναίκες με σημαντικότερα ποσοστά. Λοιπόν, κάθε τροπολογιών είναι η 6 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι. Εάν ε, δεν επιθυμεί κάποιο να λάβει το λόγο, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή και σα ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια που ακούσαμε. Χαίρομαι που αντιλαμβάνεις πως πρόκειται για μια σημαντική έκθεση και πως αυτή μπορεί να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω με τις ε, σύμβολές σας. Ε, η συμμετοχή των γυναικών θα πρέπει να τονιστεί περαιτέρω. Υπάρχουν μια σειρά κειμένων τα οποία αναφέρθηκαν και από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε πολλά στοιχεία. Ένα μια σημαντική πτυχή, μάλλον ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε, είναι ο αριθμός των χαρακτήρων, ε, αν το εκτενές ε, της έκθεσης. Ε, δυστυχώς χρειάζεται να κάνω περικοπές. Θα προτιμούσα να είχα στη διάθεσή μου πολλές, πολύ σελίδες ε, και στα εκτιμώντας θα ήθελα να καταστώ πιο αναλυτικός αλλά υπάρχει ένας περιορισμός 10.500 ε, χαρακτήρων. Εντάξει, προσβλέπω στις ε, τροπολογίες σας. Φυσικά μπορούμε και να βελτιώσουμε την έκθεση. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε κάποιες επιπλέον ιδέες. Περιμένω λοιπόν να λάβω τα σχόλιά σας και να τα συζητήσουμε. και στην τελική ψηφοφορία φαντάζομαι το κείμενο θα είναι πολύ σαφέστερο. Και τέλος, να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για όλη τη βοήθειά της. Ευχαριστώ όλους όσοι συνεργάστηκαν στενά μαζί μου Όπως σας είπα, προβλέπω στις ε, τροπολογίες σας ε, προκειμένου να βελτιώσω ακόμα περισσότερο την έκθεση. Με ευχαριστώ και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην κοινή μας ε, συνεδρίαση. Ένα λεπτό διακοπή και θα συνεχίσουμε με την κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών.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 Good afternoon everybody. Could you please take... Παρακαλώ πολύ να λάβετε τις θέσεις σας, λέει ο Πρόεδρος, για να μπορέσουμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. I, I need. Once again, please, could you take, could you take a seat, please? Παρακαλώ να λάβετε τις θέσεις σας για να περάσουμε στην ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος. Yeah. And I think it's difficult Παρακαλώ καθίστε για να περάσουμε στην ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος. Uh, Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε τώρα. Καλώς ήρθαν όλα τα μέλη των δύο επιτροπών. Είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία αυτή και σημαντική ψηφοφορία. Δυστυχώς δεν έχουμε πίνακες εδώ που προβάλλονται τα αποτελέσματα, αλλά θα τα δείτε στις μικρές οθόνες που έχετε μπροστά σας όταν θα ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Δεν έχω την κάρτα για ψηφοφορίες. Ε, εκπροσωπώ την σοσιαλιστική ομάδα και δεν έχω την κάρτα μου. Καλά, θα μετράμε την ε, ψήφο σας εδώ. Θα τη λαμβάνουμε υπόψη. Uh, το πρώτο θέμα είναι η έγκριση της ημερήσιας ε, διάταξης. Μπορούμε λοιπόν να την εγκρίνουμε. Το δεύτερο θέμα είναι το δύο ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις, άρα περνούμε κατευθείαν στην διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ε, πρόκειται για μια ψηφοφορία ανατολισμού, σημαντική Ευχαριστώ για τη συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών. Γνωρίζω ότι οι συγκητές έκαναν θαυμάσια δουλειά για να ανεβρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις. Σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Και θέλουμε να καλωσορίσουμε την κυρία Εύεριν Λέγκλερ, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Και αν θέλετε μπορείτε να λάβετε και το λόγο. Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε αμέσως την ψηφοφορία. Ωραία, όλοι πεινάνε γι' αυτό βέβαια. Η κυρία Παρβάνοβα θέλει να λάβει το λόγο. Όχι, ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω αμφότερες τις επιτροπές και τα μέλη που κατέθεσαν τροπολογίες και τους κοιόδες συγητές για την καρποφόρα στην συνεργασία αλλά επίσης και την συν ε, και λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε σύμφωνοι με τη βασική φιλοσοφία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε μέσω στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής θέλει να λάβει το λόγο, ο συνεισηγητής όχι. Ωραία λοιπόν, μπορούμε να αρχίσουμε. Αν προχωρήσω πολύ γρήγορα, μη διστάσετε να με σταματήσετε. Η ε, λίστα ψηφοφορίας έχει κάποιες παγίδες. Γιατί βεβαίως ε, όταν συμβαίνει κάτι μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη σε κάποιες άλλες τροπολογίες. Απλώς να ελέγχετε όλοι ότι είμαστε στο δρόμο. Δύο τροπολογίες, 26 και 22. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, είναι ταυτόσιμες. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική υπαριθμόν 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 24 λίμπε υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δηλαδή 28 καταπίπτει. Α, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την, την 24 της Λίμπε. Ωραία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 24 της Λίμπε. Άρχεται η ψηφοφορία. Okay. Uh, the vote is closed. Πέρας της πληροφορία. εγκρίνεται. Συνεπώς η τροπολογία 28 καταπίπτει. Περνούμε στη συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 31 και της λίμπε 27 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές δεκτή τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή η Λίμπη 28 καταπίπτει τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τούτο σημαίνει οι 76 και λείπει 29 καταπίπτουν. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 77. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is closed. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 39 τώρα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 33 της ΛΥΠΕ καταπίπτει. ΛΥΠΕ 34 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 41 καταπίπτει. Τώρα ψηφίζουμε τη ΛΥΠΕ 35. Α, είναι προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση. Ωραία, μπορούμε να ψηφίσουμε. Την ΛΥΠΕ 35. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η Λίμπε 36 καταπίπτει. Τροπολογία 79 θα ψηφίσουμε μερικός. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 80. Άρχεται ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 81 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή 83 υπέρ κατά αποχές δεκτή 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άρα η Λίμπε 37 καταπίπτει. Λίμπε 38 υπέρ κατά άποχες δεκτή. Λίμπε 39 υπέρ κατά άποχες δεκτή. Ελέγχουμε τη Λίμπε 39 άρχιτη ψηφοφορία. And the vote is closed. της ψηφοφορίας. Δεκτή. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Η τροπολογία 85 και η Λίμπε 41 καταπίπτουν. Περνούμε στη Λίμπε 42. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή οι λίμπες 43 και 44 καταπίπτουν τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή η λίμπε 45 καταπίπτει τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή λίμπε 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή και η λίπε 47 πίπτη. Και περνούμε στην 51. Τροπολογία 51. Περνούμε, ε, ψηφίζουμε μόνο τμήμα αυτής. Α, όχι, θα ψηφίσουμε το σύνολο γιατί 47. Ωραία. Υπέρ παρακαλώ της 51. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η Λίμπη 48 καταπίπτει. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η Λίμπε 40 καταπίπτει. Τροπολογία 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Λίμπε 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 55. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 56. Υπέρ. Α, ζητώ συγγνώμη. Δικό μου σφάλμα έπρεπε να ψηφίσουμε την τροπολογία ρυθμών η 55. Τώρα πάμε στην 56. Είναι προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση? Όχι, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ψηφίζουμε την 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άρα η 87 καταπίπτει. Τροπολογία 86 Ξεχωριστή ψηφοφορία σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η λίμπε 50, υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να τσεκάρουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την ΛΥΜΠΕ 50 παρακαλώ. So everybody voted. The vote is now closed. Πέρας της ψηφοφορίας δεκτή. Favor. Τροπολογία 88 υπέρ κατά εγκρίνεται. 57 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική εννέα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε στο λίμπε 52. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 53. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 54. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Yeah. 55 and Liebe 56 falls. So we then go to... 55-56 ε, καταπίπτουν. Συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να περάσουμε τώρα στην τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λίμπε 2 υπέρ. Όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ναι, τροπολογία 2 και λίμπε 2. Είναι πανομοιότυπα. Λοιπόν, περνάμε στο 22, τροπολογία 22. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 καταπίπτει. Τροπολογία 3, 3 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 και λίμπε 3, πανομοιότυπα. Θα ψηφίζουμε μαζί. Ποιοι είναι υπέρ, σηκώστε τα χέρια σα Κατά. απόχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στην τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το Λίμπε 5 πίπτη. ερχόμαστε στην τροπολογία 9, ποιοι είναι υπέρ, κατά. Όχι, με συγχωρείτε. Ναι, όχι, είναι προφορική τροπολογία. Τροπολογία προφορική. Ε, όχι, δεν θα την ψηφίσουμε. Λοιπόν, ναι, θα ψηφίσουμε υπέρ. Ε, το 62 τώρα, τροπολογία 62, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, Α το επαληθεύσουμε το 62. Αρχίζει η ψηφοφορία και την τροπολογία 62. The vote is closed. Κλείνει. Απορρίπτεται. Λίμπε 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λίμπε 7 και τροπολογία 11 μαζί είναι πανομοιότυπα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 12 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το λίμπε 8 καταπίπτει. Και το 9 καταπίπτει. Και η λίμπε 10. Τι γίνεται. Και εκείνη καταπίπτει. Και η λίμπε 13 καταπίπτει. Ερχόμαστε τώρα στην λίμπε 14. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τρία, Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 και λίμπε 12, ίδια, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε μέρος της τροπολογίας 64. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 και λίμπη 19 πανομοιότυπα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, εγκρίνονται. Λίμπη 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Το λίμπη 15 καταπίπτει. Θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να επαληθεύσουμε τη ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία για το 15, τροπολογία 15. Ψηφίσατε όλοι. Κλείνει. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 17 καταπίπτει, τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 18 καταπίπτει, συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, θα ψηφίσουμε μέρος της τροπολογίας 20. Με συγχωρείτε, λάθος. Καταπίπτει, καταπίπτει. Συνεπώς, φτάνουμε ε, στην τροπολογία 19, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβιβαστική 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, Τροπολογία 23. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24 και 21 είναι πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρο, ε, προφορική τροπολογία. Συμφωνείτε, υπάρχει αντίρρηση, όχι. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Υπάρχει αντίρρηση υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να επαληθεύσουμε αυτή την προφορική τροπολογία. Αρχίζει η ψηφοφορία για την, για την προφορική τροπολογία. Ψηφίσαν όλοι. Ψηφίσαν όλοι. Κλείνει. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 69 είναι ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτα θα ψηφίσουμε το πρώτο μέρος, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Θα πρέπει να επαληθεύσουμε πάλι την ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος αρχίζουμε. Κλείνει. Εγκρίνεται. Τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος. Κάτι είπε η κυρία. Αλλά ε, ε, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία, απορρίπτεται. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία, λέει ο πρόεδρο. Όχι, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Εγκρίθηκε, δεν απορρίφθηκε. Τώρα, το δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τώρα, όλο το κείμενο ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε, αρχίζει η ψηφοφορία. Vote Δύο λεπτά. Πρωτού φτάσουμε στην τελική ψηφοφορία. Υπάρχει κάποια σύγχυση, νομίζω, και για το ΛΥΜΠΕ 15 και την τροπολογία 15. Τι ψηφίσαμε ακριβώς, μπορείτε να μου πείτε. Θέλω να μου διευκρινίσετε τι ψηφίζαμε τελικά. Να είμαι βέβαιος ότι δεν έκανα λάθος. τρο... ψηφίσαμε την τροπολογία 15. 15. Την τροπολογία 15 ψηφίσαμε. Uh, Καλό, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε να επαναληφθεί αυτή η ψηφοφορία. Διότι ε, ψηφίζαμε σκεπτόμενοι ότι ψηφίζουμε το ΛΥΜΠΕ 15 και όχι την τροπολογία 15. Υπήρχε κάποια σύγχυση. Μήπως μπορεί να επαναληφθεί η ψηφοφορία για το 15. Το ΛΥΜΠΕ 11 απερίφθη. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Ναι, νομίζαμε ότι ψηφίσαμε το ΛΥΜΠΕ 15, ενώ ψηφίσαμε για την τροπολογία 15. Συμφωνείτε, ναι, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 15. Είναι η καλύτερη μέθοδος. Λοιπόν, το βρήκατε στη σελίδα 9. Τροπολογία 15. Ξαναψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Καταλάβατε τώρα τι ψηφίζουμε. Πολύ, πολύ καλά. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 15. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τελειώσατε. Κλείνει. Νομίζω ότι εγκρίθηκε τώρα. Εντάξει, εντάξει, όχι. Είναι προτιμότερο να κάνει κανείς διπλό έλεγχο. Τώρα, η τελική ψηφοφορία για το σύνολο για όλο το ψήφισμα. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Τώρα αρχίζει για όλο το κείμενο. And the vote is closed. Κλείνει. Με, ε, χωρίς ε, αμφισβήτηση εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Thank you very much everybody. Ευχαριστώ πολύ. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ.